starting the Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Παρακαλώ, θα ελέγξουμε λειτουργεί το σύστημα. Γι' αυτό αν έχετε την καλοσύνη, ε, βάλτε τις κάρτες σας στο μηχάνημα για να το δοκιμάσουμε. Θα γίνει έλεγχος του συστήματος ψηφοφορίες. Παρακαλώ ψηφίστε για να δούμε αν λειτουργεί πάλι τις κάρτες σας. I'm trying to make... So I have... I forgot the card in one, two minutes. Έχω ξεχάσει την κάρτα μου. Σε ένα-δύο λεπτά θα καταθέσει βοηθός με την κάρτα. Αλλά στο μεταξύ θα ψηφίζω με το χέρι. Okay. There are two cards in the machines which were και έχουμε και μια κάρτα που φαίνεται να μην λειτουργεί μέσα στο μηχάνημα. Ψηφίζουμε πρώτα το σχέδιο γνωμοδότησης. Καταρχήν ποιο είναι πρώτο να δούμε. είναι σχέδιο κανονισμού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τη μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδιότητα εκδικάσεω σε πρώτο βαθμό των διαφορών μεταξύ τη Ένωση και των υπαλλήλων Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται, δεν χρειάζεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Which means that the judges will have... Άρα, ε, όσοι ψήφισαν κατά, ε, προτιμούν να έχουμε δικαστές που θα μένουν με σταυρωμένα τα χέρια, γιατί αυτό σημαίνει, θα μεταταχθούν οι δικαστές για να αναλάβουν στο Γενικό Δικαστήριο. Πάμε στην ετήσια έκθεση του 2004 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Συμβαστική τροπολογία Α, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται, η 7 έχει αποσυρθεί. Πάμε στην 12, ποιος είναι υπέρ. Τροπολογία 12, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 κατά πίπτη. Πάμε στη βασική τροπολογία Β, ποιος είναι υπέρ. Κατά τμήματα, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται. Πάμε στην 23, ποιος είναι υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία C ποιο είναι υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική τροπολογία C. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Με μία ψηφοδιαφορά, αλλά εγκρίνεται. 28, ποιος είναι υπέρ, τροπολογία 28. 8 28 σοσιαλιστές κατά ηλεκτρονικός έλεγχος αν και κατά τη γνώμη μου έχει εγκριθεί. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται όντως. Πάμε στην τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ? 28 εγκριθήκε. 15 προς 7 και μία εποχή. 30. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 8 προς 15 κατά. Θα το διαβάζω γιατί νόμιζα το βλέπατε και εσείς στις οθόνες, αλλά φαίνεται ότι δεν εμφανίζεται. «8 υπέρ 15 κατά απορρίπτεται». «38 ποιος είναι υπέρ» κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία δέλτα, D. 9. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 40. Πέντε τροπολογία, αλλά για το δεύτερο τμήμα μόνο. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, μάλλον εγκρίνεται έτσι. 46, Ποιο είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 46, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 6 υπέρ, 16 κατά και μία αποχή. Απορρίπτεται. Πάμε στην 50. Τροπολογία ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ε. Υπέρ. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Για το δεύτερο τμήμα, ποιο είναι υπέρ. Δεύτερο τμήμα τη συμβαστική ε, Ποιο είναι υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62 τροπολογία, ποιος είναι υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ας το ελέγξουμε. 64. Τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται με 5 ψήφους υπέρ 15 κατά και 3 αποχές. Περνάμε στην 65 κατά αποχές απορρίπτεται και η τελευταία τροπολογία 66 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τελική ψηφοφορία της γνωμοδότησης. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 22 υπέρ, μία ψήφος κατά, χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια. Θετικό το αποτέλεσμα. Κύριε Ουγιασδόφσκι. Και πάμε σε αφήσει από το πρωί το σημείο 6, την προετοιμασία δηλαδή της μετακλογικής αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, για να δώσουμε την συνεισφορά μας πριν υποβάλει την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Πέντρο Σίλβα Περέιρα εκπώνησε τη γνωμοδότηση. Έχει το λόγο, Πέντρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε σύντομα σχόλια μόνο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που κατέθεσαν. Οι περισσότερες εκ των οποίων παρέσχουν μια πολύ σημαντική, πολύ επικοδομητική συνεισφορά ως παρέμβαση. Με βεβαιότητα μπορούν να βελτιώσουν το κείμενο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια θέματα εν τούτης, το πρώτο από αυτά είναι ότι για την ίδια την ιδέα ότι φυσικά αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα νέες τεράστιες προκλήσεις εξειδικευμένα πρέπει να αναφέρουμε ξεχωριστά την προσφυγική κρίση ως πρόκληση επίσης ε, την τρομοκρατική απειλή και τις ε, διακούσες πτυχές της οικονομικής ε, κρίσης. Όλοι αυτοί οι συντελεστές θα απαιτήσουν μεγαλύτερη ελαστικότητα, μεγαλύτερη ευλήγησία όσον αφορά τους κανόνες και κανονισμούς για τα δημοσιονομικά και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αναθεώρηση των πολιετών δημοσιονομικών πλαισίων. Με την αναθεώρηση εννοούμε φυσικά πιθανότατα ή δυνατόν μια αύξηση των κονδυλίων σε σχέση με τα πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια που θα τεθούν υπό συζήτηση έγκριση. Λοιπόν, και να επικεντρωθούμε επίσης ε, στα υφιστάμενα ανώφλια των ε, ενισχύ πολιετών δημοσιονομικών πλαισίων για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Να γνωρίζουμε όμως με αφήνει ότι οποιαδήποτε αύξηση ελαστικότητας στην κατανομή κονδυλίων πρέπει να βαίνει εκ παραλίλου με μια ισχυρότερη ε, πτυχή οικονομικού ελέγχου ε, από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης αναφέρεται και η ανάγκη να υπάρξει ενότητα του προϋπολογισμού σε ένα ενιαίο πλαίσιο μέσα στα πλαίσια της ε, λογοδοσίας και της διαφάνειας όσον αφορά τις τελικές ε, αποφάσεις και ένα προϋπολογισμό που θα βρίσκεται ε, στο ύψος των αναγκών δημοσιονομικά. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τους ιδίους πόρους, η προσέγγιση μου φυσικά είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα στην ίδια άσκηση, στο ίδιο εγχείρημα το οποίο παρακολουθούμε ξεχωριστά, εδώ δεν νομίζω ότι είναι ίσως τη θέση να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες σε όλα αυτά τα θέματα και γι' αυτό απλά και μόνο μια ισχυρή στεναρή δέσμευση για την δημιουργία ενός ε, πλαισίου ιδίων πόρων που θα είναι αποφασιστική σημασίας και που θα πρέπει αυτό να εξεταστεί υπό τις πρωτοβουλίες που συζητήθηκαν σήμερα το πρωί όσον αφορά τα θέματα του Παύλου Ραντζέο. Γενικά θα έλεγα ότι με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί μπορούμε να καταλήξουμε σε εύθετους σκόπιμους συμβιβασμούς και θα έχουμε και μια συνάντηση σχεδόν εισηγητών το δυνατόν πιο ε, νωρίς, πιο γοργά για αυτό. Σας ευχαριστώ όλους σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σκιώθησε για το ΕΛΚΑ, ο κύριος Σεπφλίν, Γιώργη Σεπφλίν. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τα προαναφερθέντα. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό να γίνει και συμφωνώ. <clears throat> Κανείς δεν θα αμφισβητούσε ότι αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις μεγάλης εμβέλειας και όλα αυτά για τα οποία γίνεται λόγος εδώ πρέπει να αντανακλούν αυτές, την απέτηση να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Θέματα όπως οι πρόσφυγες, η τρομοκρατία, η οικονομία κτλ. Τώρα για την ελαστικότητα, σωστό είναι αυτό νομίζω, ούτε δεν είναι καθόλου εύκολο το εγχείρημα να διαρθρωθούν όλα αυτά όταν κάνουμε λόγο εξελίξεων όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα ότι οι ήδη πόροι θα έπρεπε να ε, μην έχουν την ανώτατη προτεραιότητα. παρόλα αυτά θα πρέπει να το συζητήσουμε και αυτό στην διεξαγωγή μια συζήτηση σε ευρύτερα πλαίσια ώστε να αντανακλώνται οι προοπτικές της ε, ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης. Σας ευχαριστώ λοιπόν και με αυτές τις τροπολογίες πάμε καλά, βαίνουμε καλώς. Ευχαριστώ. So the other Οι άλλοι σκιώδεις, ο κύριος Γκιόρενς από την Άλντε ίσως. Δεν παρίσταται, ωραία. Πασκάλ ε, Ντυρόν, Κάποιος από τους πράσινους, όχι. Μάσιμο Καστάλτο ήταν εδώ προηγούμενα. Άλλοι. Κύριε Σογιασδόφσκι. Θα ήθελα να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα τα πολωνικά. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Περέιρα για την ε, εκπόνηση της γνωμοδότησής του. Πιστεύω ότι για το θέμα αυτό θα πρέπει να μεριμνήσουμε πρώτα απ' όλα για τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και είναι αλήθεια ότι η οικονομική και η δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί ελαστικότητα. Απαιτούν ε, ευελιξία προκειμένου να προσαρμοστούμε και να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες ε, προκλήσεις ε, που μας περιέγραψε ο κύριος Περέιρα, το προσφυγικό, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό γίνεται πιο συγκεκριμένο, ακριβές και σταθερό. Και εγώ, όπως και ο κύριος Σέπλιν, θα ήμουν υπέρ ε, του να διεκπαιρεώσουμε αυτό το θέμα ε, της, των ιδίων πόρων. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της σταθερότητας και της ευελιξίας που χρειάζεται, καθώς και των διορθώσεων στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και ευχαριστώ τον κύριο Περέιρα και είμαι έτοιμος για περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Μπρέσο. Εφόσον τελειώσαμε με τους πιο δυσηγητές, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συντάκτη της γνωμοδότησης για την γνωμοδότησή του αυτή, που είναι ευσύνοπτη βέβαια γιατί υπάρχουν οι πολύ συγκεκριμένοι κανόνες για την έκταση των γνωμοδοτήσεων όπως το γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά καταφέρνετε πραγματικά να επικεντρωθείτε στα βασικά σημεία που θα πρέπει να μας απασχολήσουν στα πλαίσια της αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και μάλιστα κάνετε και κάποιες περαιτέρω προτάσεις. Η φυστάμενη αυτή μάλλον η μελλοντική αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να συμπεριλάβει σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον τους ίδιους πόρους. Ούτε νομίζω ότι θα καταφέρουμε να αυξήσουμε τα ανώτατα όρια, αλλά μη τι άλλο μπορούμε να διευθετήσουμε το ζήτημα της ευελιξίας και ενδεχομένω της ευθυγράμμισης των πιστώσεων πληρωμών βάσει των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα σε αυτά τα δύο δεδομένα που δημιουργεί τελικά πάρα πολλά ποσά τα οποία οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία δεν έχει καταβάλει. Στη γνωμοδότηση αυτή μας δίνονται και κάποιες ενδείξεις για το πώς θα μπορούσαμε ακόμα και στα πλαίσια αυτής της επόμενης αναθεώρησης να κάνουμε κάποιες δεσμεύσεις για το μέλλον, για το απότερο μέλλον, ιδίως όσον αφορά τους ιδίους πόρους, ιδίως όσον αφορά ένα προπολογισμό για την Ευρωζώνη, και ενδεχομένως ακριβώς αυτό το τελευταίο ζήτημα, με την καλή θέληση βέβαια και τη βοήθεια των κρατών μελών, θα μπορούσε να ελοποιηθεί ακόμα και στην ε, ενδιάμεση αυτή φάση της αναθεώρησης. Γιατί υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ζήτησε αξιολόγηση, αλλά αναθεώρηση. Αναθεώρηση μπορεί να συνεπάγεται ακόμα και τροποποίηση των συστατικών στοιχείων του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Έτσι λοιπόν, επεξεργαζόμενος ο συντάκτης γνωμοδότης τροπολογίες θα μπορούσε να τονίσει εκ νέου την έκκληση αυτή που είχε κάνει στο παρελθόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί θα αποτελέσει σίγουρα πολύ σημαντικό στοιχείο της όλης διαδικασίας αναθεώρησης που θέλουμε, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα περιοριστούν σε μια πολύ ελαφριά αξιολόγηση τα κράτη-μέλη, χωρίς να επιφέρουν σημαντικές προσαρμογές ή σημαντικές τροποποίησεις χωρίς δηλαδή να καταφέρουν να εξασφαλίσουν περισσότερους πόρους για τις τόσες πολλές δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει στο παρελθόν το Συμβούλιο και που συνεχίζει και παίρνει βέβαια, ιδίως όσον αφορά το προσφυγικό ζήτημα, όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας και της προστασίας, όσον αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο ακτοφυλακής και συνοριοφυλακής, για όλες αυτές τις πολιτικές πρωτοβουλίες απαιτούνται περισσότεροι πόροι και δεν θα πρέπει προφανώς αυτοί να αντληθούν από την κοινή γεωργική πολιτική, από την πολιτική συνοχής. Πρέπει λοιπόν να μας πει το Συμβούλιο από πού θα προέλθουν οι πόροι αυτοί. Νομίζω λοιπόν ότι και το ζήτημα αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στα βασικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν στα πλαίσια της Αξιολόγηση και αναθεώρησης του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε Μερτσέντε. Άλλοι ομιλητέ, ο κύριο Περέρα, ο στάκτης νομοδότης, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μια τελική παρατήρηση απλώς για να ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις που έγιναν και να υπογραμμίσω ότι αυτό περί του οποίου πρόκειται στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού πολιτικού πλαισίου είναι μεγάλη σημασία, είναι πραγματικά μεγάλη σπουδαιότητα. Σε μια χρονική στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις, αυτές τις τεράστιες προκλήσεις, πραγματικά το να ξαναδεί κανείς τα μέσα που θα έχει στη διάθεσή της αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η λιδία λίθος για την ίδια την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την πολιτική βούληση που πρέπει να υπάρχει για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Και έχουμε εδώ και σε σχέση με αυτό το εγχείρημα στην ε, διάρθρωση, οικοδόμηση αυτού του αρχικού δημοσιονομικού πλαισίου και που οδήγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαιτήσει τη διαδικασία εμβαθυμένη αναθεώρησης που είναι αυτό το οποίο θα αναπτύξουμε τώρα ως εγχείρημα. Το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι σε μια στιγμή όπου επιδεινώνονται τα προβλήματα ακόμα περισσότερο όσον αφορά την τοποθέτηση των ίδιων των Ευρωπαίων πολιτών να μην είναι σε θέση να δώσει απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη συγκυρία. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων και για την διαθεσιμότητα κονδυλίων από πλευράς των μέσων των δημοσιονομικών να διεξαχθεί και μια συζήτηση για τα μέσα και εργαλεία ελαστικότητας του δημοσιονομικού πλαισίου για να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει και για να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό διασφαλίζοντας την σταθερότητα και την ισορροπία όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι για την επίτευξη κυρίως των μιζώνων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της συνοχής με αυτή την προσαρμογή κονδυλίων, τον επιμερισμό κονδυλίων στους νέους ε, προκλήσεις, στις νέες προκλήσεις, να μην γίνουν θυσίες, να μην υπάρξουν περικοπές, πράγμα το οποίο είναι και αυτό σημαντικό σε αυτή τη χρονική στιγμή για την ε, συνοχή. Αυτή είναι η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ενώπιόν μας. Θα συνεργαστούμε από κοινού τις δικές σας και πιστεύω και ευελπιστώ ότι στη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών που πολύ σύντομα, πολύ γοργά θα διεξαρθεί, θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε προτάσεις που θα είναι πραγματικά επικοδομητικές. Ευχαριστώ. Ε, Εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο, τότε ας περάσουμε στο διάταξης ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 29 Οκτωβρίου του 2015, ο κύριος Ραμόν Ιαρέγκια Τόντο διορίστηκε εισηγητής έκθεση ιδίες πρωτοβουλία όσον αφορά την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνατότητες και προκλήσεις, η Επιτροπή Πολιτισμού και συγκεκριμένα η κυρία Ζαμπέλα Ντινόλφη εξ ονόματο της Επιτροπής αυτής θα γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια τη της προηγούμενης συνεδρίας της Επιτροπής μας στις 14 Μαρτίου η Επιτροπή μας διοργάνωσε μια δημόσια ακρόαση για το ζήτημα αυτό τη ηλεκτρονική δημοκρατία λέγοντας ότι όντως φέτος θέλουμε να επικεντρωθούμε σε νέους καινοτόμους, καινοτόμες μορφές δημοκρατίας και θέλαμε να δούμε πώς μπορούμε και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλουμε στη νέα αυτή διαδικασία, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, στην πολιτική ζωή, προκειμένου να επαναφέρουμε τους πολίτες ε, πίσω στην δημόσια αυτή ε, δραστήρια ενασχόληση με την πολιτική. Το άρθρο 11 της συνθήκης λέει ξεκάθαρα ότι τα θεσμικά όργανα και παραθέτω μέσω των κατάλληλων μέσων θα δώσουν στους πολίτες και στις, στους οργανισμούς εκπροσώπησης των πολιτών την δυνατότητα να γνωστοποιούν τις απόψεις τους σε όλους τους τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε περισσότερο την ψηφιακή τεχνολογία προκειμένου να ενισχύσουμε την συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να δώσω τον λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Αουρέγγι, ο οποίος θα μας παρουσιάσει καταρχάς ένα έγγραφο εργασίας για το ζήτημα αυτό. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα στους αγαπητούς συναδέλφους ότι η συζήτηση για την ηλεκτρονική δημοκρατία, το e-democracy, Ε, είναι πολύ ευρύ, παρά είναι γενικό και αόριστο. Γι' αυτό θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε περί τίνος πρόκειται και τι πράγμα μιλάμε. Το θέμα της ηλεκτρονικής δημοκρατίας είναι πολύ σημαντικό και αποτελεί και αντικείμενο μελετών σε πάρα πολλά πανεπιστήμια του κόσμου. Σε πολλές χώρες ε, έχουμε συγκεκριμένες πρακτικές και θα μπορούσαμε κάλλιστα ε, επί τη ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε και εμείς εκτενέστατες μελέτες, αλλά καλό θα ήταν να συγκεκριμενοποιήσουμε εδώ και να περιορίσουμε το πεδίο της ε, έκθεσης μας. Η προσέγγιση μου είναι εξή. Η δημοκρατία, το ισχύο σύστημα ε, συμβίωσης ε, και ελευθερίας δεν πάει καλά. Οι λόγοι για την λεγόμενη δημοκρατική κρίση, ή την απαξίωση των θεσμών, ή την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ πολιτικού κόσμου και πολιτών. Επίσης είναι θέμα πολυάριθμων μελετών, ερευνών και βιβλίων. Πάντως, χονδρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται την πολιτική ως κάτι ξένο, και περίπλοκο και είναι όλο και πιο δύσκολο να εξηγήσουμε στους συμπολίτε μας τις αποφάσεις μας και είναι και δύσκολο για τους συμπολίτε μας να κατανοήσουν αυτές τις αποφάσεις, πολλές από αυτές. Και ιδιαίτερα στα οικονομικά θέματα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές περιορίζουν κάπως την άσκηση της άμεσης δημοκρατίας. Υπάρχει πρόβλημα και με την παγκοσμιοποίηση, γιατί η παγκοσμιοποίηση περιορίζει το δημοκρατικό πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις. Ο Ρόντρικ, ε, ο στοχαστής, ε, ο θεωρητικός, είναι αυτός που ε, ε, μελέτησε καλύτερα αυτό το καταραμένο τρίγωνο μεταξύ κράτους, παγκοσμιοποίησης και δημοκρατίας. Κατά λίγο το συμπέρασμα ότι όσο, δυνατό περισσότερη, όσο περισσότερη παγκοσμιοποίηση έχουμε, τόσο λιγότερη δημοκρατία έχουμε. Επίσης έχουμε και μία ρήξη του κοινωνικού συμβολέου. Ε, από την άποψη ότι όλο και περισσότεροι πολίτες ε, δεν βλέπουν το κράτος ως κράτος προστάτη αλλά με την κρίση αισθάνονται όλο και πιο ανήμπεροι και όλο και πιο ανυπεράσπιστοι από πλευράς του κράτους και αυτό τους απομακρύνει ακόμη περισσότερο από την πολιτική και τον πολιτικό κόσμο. Οπότε η πρώτη διαπίστωση είναι ότι η δημοκρατία δεν πάει καλά. Δεύτερη διαπίστωση. Στην τεχνολογία, στα δίκτυα, στις, στους νέους μηχανισμούς επικοινωνίας στα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social media, τι υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να διευκολύνει και να βελτιώνει τη δημοκρατία, που όπως είπαμε δεν πάει καλά. Η έκθεση προσπαθεί να βελτιώσει τη δημοκρατία ή να λύσει αυτά τα προβλήματα ε, τότε το ερώτημα αν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο και να το αξιοποιήσουμε καλύτερα για να ανακτήσουμε ή να αναβιώσουμε τη σχέση μεταξύ πολιτών και πολιτικού κόσμου. Αυτή είναι η σκοπιά της έκθεσης. Ε, περιγράφω και αναφέρω κάποιους ορισμούς από τη θεωρία για να δούμε τα διάφορα σκέλη αυτής εξίσωσης και θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ τριών ενιών. Ε, τεχνολογία και δημοκρατία είναι η μία. Έχουμε φαινο τα, μέσα κοινωνικής ε, δικτύωσης, ε, τα στιξ και βλέπουμε ότι υπάρχει μια βελτίωση στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών από πλευράς κυβερνήσεων προς τους πολίτες. Μιλούμε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση γιατί η ίδια η διακυβέρνηση υπόκειται σε νέους μηχανισμούς επικοινωνίας, ε, συμμετοχής στη συζήτηση, καλύτερης ενημέρωσης, περισσότερης διαφάνειας, ώστε οι αποφάσεις ε, των πολιτικών ηθινών στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να έρχονται πιο κοντά στους πολίτες. Και μιλούμε και για ηλεκτρονική δημοκρατία, δηλαδή στη χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, προκειμένου να δημιουργήσουμε διάβλους επικοινωνίας, ε, για την αμυγή πολιτική δράση. Ε, εκλογές με ηλεκτρονική ψήφο, την ηλεκτρονική βουλή, την ηλεκτρονική πρωτοβουλία, διαβουλεύσεις μέσω του διαδικτύου. Οπότε έτσι έχουμε μια πιο έντονη δημοκρατία χάρη στη χρησιμοποίηση των δικτύων. Σε μια άλλη παράγραφο κάνω μια ε, απεικόνιση της κατάστασης. Λέμε σε τι φάση βρισκόμαστε. Μάλιστα αναφέρω τα, τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάποιων μεμονωμένων χωρών. Ε, περιγράφω δηλαδή τις βέλτιστες πρακτικές, ε, κάποιες ενδιαφέρουσες εμπειρίες που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε στο μέλλον για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό της ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Σε ένα άλλο κεφάλαιο αναφέρω τους δυνητικούς κινδύνους μίας διεύρυνσης της ιδέας που δεν λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα της εφαρμογής της. Στο σχέδιο της έκθεσης που σας υποβάλλω επισημαίνω πέντε μείζωνα προβλήματα που δεν μπορούμε να παραγωνίζουμε. Για παράδειγμα, το ψηφιακό χάσμα, όχι μόνο το υλικό, λόγω της έλλειψης πρόσβασης στο ίντερνετ σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά και το χάσμα ε, λόγω της, του ψηφιακού αναλφαβητισμού. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που δεν είναι εξοικειωμένος με αυτές τις τεχνολογίες και δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτά τα δίκτυα. Υπάρχει και το θέμα της, εκλογικής απάτης, αν έχουμε ηλεκτρονικά συστήματα ψηφοφορίας. Επίσης, έχουμε το θέμα της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας και των προσωπικών δεδομένων. Και αυτά είναι, ένα στοιχείο, ε, και αυτά είναι στοιχεία προ εξέταση. Και τέταρτον, ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Το δίκτυο είναι ο ιδανικός χώρος για τη συζήτηση. Δηλαδή, το διαδίκτυο, γενικώ τα δίκτυα μπορούν να, να ενισχύσουν ε, τη, σε βάθος την κριτική σκέψη. Ή μήπως ε, ε αναδεικνύουν περισσότερο ακραίες ε, ε, ή μειονοτικές απόψεις. Επίσης, όσο μεγαλύτερη διαφάνεια έχουμε και όσο περισσότερο μιλούμε για την διακυβέρνηση, η χρήση αυτών των εργαλείων, των μηχανισμών, των τεχνολογιών και της πληροφορίας μερικές φορές γίνεται μονοπόλιο όχι των πολιτών αλλά συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων που χρησιμοποιούν αυτές τις ευκαιρίες για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα ή τα συντεχνιακά συμφέροντα. Και δυστυχώς αυτό βλέπουμε από τις εμπειρίες μας. Αυτά τα συμφέροντα και οι ομάδες συμφερόντων χρησιμοποιούν περισσότερο τα δίκτυα. Και ολοκληρώνω την έκθεση με αναφορά της ακολουθητέας πορείας και απαρίθμηση κάποιων στοιχείων και κάποιων προτάσεων. Δηλαδή, αναφέρω 7 κατηγορίες με αντίστοιχες πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην πολιτική. Για παράδειγμα, να ενισχύσουμε την ενεργό συμμετοχή των εκπροσώπων των πολιτών στα υπάρχοντα φόρα για να προωθήσουν τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. Επίσης, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Άλλη πρωτοβουλία θα ήταν χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες να επιτρέψουμε την πρόσβαση στην πληροφορία, τη διαφάνεια και την ενεργό συμμετοχή, ηλεκτρονική διακυβέρνηση δηλαδή, δίκτυα συμμετοχής με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για να ενισχυθεί η έρευνα και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και μηχανισμών. Πέμπτον, να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι που προανέφερα ώστε η χρήση των τηλεπικοινωνιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να μην διαστρεβλώσουν την ίδια την ουσία, την πεμπτουσία της δημοκρατίας, έκτο να προωθήσουμε τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και τέλος ε, ε, δίνουμε στα πολιτικά κόμματα νέα συστήματα ανοίγματο και επαφή και επικοινωνίας με τους ε, πολίτες και τους, τα μέλη του κόμματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ξέρετε, ε, έχει περιορισμούς τους χαρακτήρες για τέ, τέτοιου είδους εκθέσεις και ευχαριστώ και τις υπηρεσίες για τη βοήθειά τους, αλλά δυστυχώς ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους περιορισμούς ως προς την έκταση του εγγράφου. Πάντως προσπαθώ να κάνω μια αυστηρή και σοβαρή περιγραφή και οριοθέτηση της πολιτικής συζήτησης. Ε, για τη δημοκρατία μας, την κρίση της και τις ευκαιρίες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες. Δεν θέλω η συζήτηση ε, να μετασχηματίσει, να μεταμορφώσει το δημοκρατικό σύστημα. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα της ε, αντι, αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Απλώς θέλουμε να το βελτιώσουμε. Και οι τεχνολογίες αυτές της επικοινωνίας αποτελούν δεν αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία που θα μεταμορφώσουν τη δημοκρατία και θα επιλύσουν ω διαμαγεία όλα τα προβλήματα που ανέφερα. Μπορούν να είναι ένα εργαλείο για να τελειοποιήσουν το δημοκρατικό μοντέλο, αλλά όχι για να αλλάξουν την ουσία τη αντιπροσωπευτική δημοκρατία που κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη μορφή δημοκρατία. Τι άλλο επιδιώκουμε. Μία αντικειμενική και ισορροπημένη περιγραφή μεταξύ του δυναμικού και των κινδύνων, των ευκαιριών και των κινδύνων, και αυτό το εξηγούμε. Και τέλο ένα οδικό χάρτη ε, στην πολιτική συζήτηση σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο και με τους διάφορους πολιτικούς τελεστές, δηλαδή τα μέσα επικοινωνίας, τα πολιτικά κόμματα και το καθεξής. Μια και είμαστε υποχρεωμένοι να περιορίσουμε σε πέντε σελίδες την έκθεση, εγώ περιμένω τις προτάσεις σας πριν εκπονήσω το προσχέδιό μου. Θα περιμένουμε και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων επιτροπών. Θα είναι πολλές αυτές που θα γνωμοδοτήσουν για το θέμα και περιμένω και από εσά τα βιώματά σας, τις εμπειρίες σας, τις προτάσεις σας και τις ιδέες σας. Γιατί παρόλο που δεν πρόκειται να αλλάξουμε τον κόσμο, πιστεύω ότι με αυτό το έγγραφο, μη τι άλλο, κάπως θα τον βελτιώσουμε. for the e Christian Από το ΕΛΚ τώρα, σχεδόν ο Κρίστιαν Dan Πρέντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. για αυτό το έγγραφο εργασίας. Θα επικεντρωθώ σε τρία σημεία. Πρώτον, η αιτιολόγηση που δίνεται όσον αφορά την αναγκαιότητα μιας τέτοιας έκθεσης. Στην αρχή μάλιστα τον γράφου σας αναφέρεστε σε αυτό. Συμφωνώ με τις διαπιστώσεις του εισηγητή, δηλαδή ότι ανάμεσα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, υπάρχει μια απαξίωση, μια παθητική στάση, μια απογοήτευση, ακόμα και μια ρίζοσπαστικοποίηση ότι πολλές φορές έχουμε διάφορες ε, περίεργες ε, ε, αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία, στο Παρίσι, που υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι περνάνε όλο το τις πλατείες της πόλης. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ε, είναι εξίσου σημαντικό να τονίσουμε κυρίως ε, τη χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές. Εκεί πέρα που ε, δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις εκλογές, στις χώρες που δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις εκλογές. Στο πρώτο τμήμα του εγγράφου αιτιολογείται γενικά την αναγκαιότητα μιας τέτοια έκθεσης. Δεν θα ήθελα να σας δυσαρεστήσω, είχα την εντύπωση ότι διάβαζα το πρόγραμμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο προήμιο της έκθεσής σας. Γιατί ξέρω ότι όλο αυτό το θέμα σας αρέσει πάρα πολύ. Ο κίνδυνος της παγκοσμιοποίησης, οι κακές χρηματοπιστωτικές αγορές, τις οποίες πρέπει να ελέγξουμε. Τι άλλο μας λέτε εδώ για να δω. Λέτε ότι περιορίζουν τις ίδιες πολιτικές αποφάσεις αυτές οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Αναφέρεστε στο σύστημα διακυβέρνησης του ευρώ. Βλέπω σιγά σιγά ότι στρέφεστε κατά διαφόρων πολιτικών και της πολιτικής λιτότητας. Εσείς έχετε τη δική σας πολιτική άποψη. Υπάρχουν άλλες πολιτικές οικογένειες, άλλες πολιτικές ομάδες που προσεγγίζουν διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν θα πρέπει στην αρχή του εγγράφου αυτού να γίνει μια τέτοια πολιτική συζήτηση και ανάλυση. Ανταυτού νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις νέες μορφές έκφρασης, στις νέες κινητοποιήσεις, στην ε, συμμετοχή όσον αφορά την πολιτική ζωή. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις σχέσεις οικονομίας και πολιτικής, άλλωστε επ' αυτού διήστανται οι απόψεις μας, αλλά Θα ήταν πιο ενδιαφέρον αντί να κάνουμε τόσε αναφορέ στην οικονομική κρίση ή στα δεινά τη παγκοσμιοποίηση ή γενικότερε επιπτώσει παγκοσμιοποίηση, να δούμε καλύτερα ποια είναι η στα δεινα τη παγκοσμιοποιηση η γενικοτερε επιπτωσει πτυχή του συστήματος αυτού που προτείνεται της ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Το πολιτικό δηλαδή αν θέλετε περιεχόμενο περισσότερο θα πρέπει να μας απασχολήσει και όχι να κάνουμε διάφορες εκτιμήσεις οι οποίες άλλωστε έχουν να κάνουν με την πολιτική κατεύθυνση την οποία ακολουθούμε. Όσον αφορά τώρα την ίδια την οριοθέτηση του ζητήματος, συμφωνώ εδώ με τον εισηγητή όταν μας λέει ότι δεν θα πρέπει εκ νέου να προβλέψουμε έναν νέο ορισμό για την ηλεκτρονική δημοκρατία και ότι είναι καλύτερο να βασιστούμε σε έναν ορισμό που έχει προτείνει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να καταφέρουμε να οριοθετήσουμε λίγο περισσότερο τον ίδιο το στόχο αυτής της έκθεσης. Επί ποιων ζητημάτων θέλουμε να επικεντρωθούμε πιο συγκεκριμένα. Στις σελίδες 3 και 4 έπειτα του εγγράφου εργασίας πολλές φορές ε, αντιμετωπίζουμε με αρκετά λεπτομεριακό τρόπο διάφορες μορφές ηλεκτρονικής δημοκρατίας όπως αυτές εμφανίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνεται διάφορα παραδείγματα όπως ε, την επιτυχία του ηλεκτρονικού συστήματος ψηφοφορία στην Εστονία. Στη συνέχεια όμως κάνετε και κάποιες αναφορές σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρεστε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και το καθεξής. Χάνουμε κάπως τη διάσταση την οποία θέλετε να φωτίσετε περισσότερο. Επικεντρώνεστε περισσότερο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στο εθνικό επίπεδο και στα δύο ενδεχομένω. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι δημιουργούμε έναν συνοθήλευμα και είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε τελικά να φωτίσουμε επακριβώς τη μία ή την άλλη πλευρά. Χαίρομαι και εγώ για την επιτυχία διαφόρων πρωτοβουλειών, όπως για παράδειγμα η πρωτοβουλία που είχαμε στην Εστονία. Άλλο να λέμε βέβαια ότι υπάρχουν κάποιες ε, ε, επιμέρους επιτυχίες ή κάποια παραδείγματα τα οποία λειτουργήσαν εδώ και εκεί θετικά και άλλο να λέμε ότι θέλουμε να εισάγουμε ένα ηλεκτρονικό εκλογικό σύστημα σαν αυτό της Εστονίας. Θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη, εφόσον θέλουν, να ακολουθήσουν το σύστημα αυτό. Εγώ θα το πρότεινα στη τελευταία ανάλυση. Τρίτη παρατήρηση στη συνέχεια. Ποιες είναι οι συστάσεις που θα διατυπώσουμε στην έκθεση αυτή. Έχουμε την πρόκληση αυτή ενώπιόν μας να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα επιτρέψουν στον πολίτη να επανασυνδεθεί με τον κόσμο της πολιτικής, να επενδύσει εκ νέου στην πολιτική, να αρχίσει να συμμετέχει περισσότερο. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι κάποιες άτακτες αντιδράσεις κατά της ίδιας της πολιτικής. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν τον πολίτη να επανασυνδεθεί με την πολιτική σκηνή, με τους πολιτικούς και δεν να χρησιμοποιώ τυχαία τον όρο επανασύνδεση, εφόσον μιλάμε άλλωστε και για ψηφιακή τεχνολογία. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα, πρέπει να καταβάλουμε γι' αυτό διάφορες προσπάθειες και έπειτα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε προγράμματα κατάρτισης ε, στις νέες τεχνολογίες, Νομίζω ότι επ' αυτού πρέπει περισσότερο να επικεντρωθούμε και να μην μπερδέψουμε πάλι πολλά διαφορετικά πράγματα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, ξεφύγουμε λίγο από τις ιδεολογικές αγκυλώσεις που μπορεί να έχει μία ή άλλη πολιτική ομάδα. Κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα και αυτή είναι η πραγματική πρόκληση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Εξ ονόματος του ECR, ο κύριος Σουζαντόφσκι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω παράπονα από τον εισηγητή επειδή εξέφρασε τις κομματικές του απόψεις. Ισχύει εδώ η πολυμορφία. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε το τελικό αποτέλεσμα, η τελική έκθεση, να είναι όσο, πιο γίνεται, όσο γίνεται πιο συγκεκριμένη. Και αυτό που θα πω είναι φυσικά η δική μου πρόταση για να οργανώσουμε μία δημόσια ακρόαση που να επικεντρώνεται ακριβώς στους νέους τρόπους και στα νέα μέσα έκφρασης πολιτικής ε, ε, θέσεις και σε συνεργασία με διάφορα πανεπιστήμια. Νομίζω ότι έτσι θα εμπλουτίσουμε την έκθεση και θα βοηθηθούμε για να μπορέσουμε να συντάξουμε μια τεκμηριωμένη έκθεση για την ηλεκτρονική δημοκρατία. Θα ήθελα λοιπόν επ' ευκαιρία τη εκπόνηση αυτή τη έκθεση να οργανώσουμε δημόσια κρόση με εμπειρογνώμονε, πανεπιστημιακού, επιστήμονε που ασχολούνται ειδικά με το θέμα των νέων μορφών συμμετοχή και νέων μορφών πολιτική έκφραση στο διαδίκτυο. Αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα μα βοηθήσει όλου μια τέτοια δημόσια κρόση. Ευχαριστώ. Η Μάιτα, δεν κάνω λάθο, θα μιλήσει για την άλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε με ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο που παρουσίασε ο εισηγητής είμαι Ισπανίδα. Έχω λιγότερη απόσταση πολιτισμική ε, όσον αφορά αυτά τα θέματα σε σχέση με τον εισηγητή και από τους ε, Ισουίτες και μου φαίνεται ουσιαστικό να παρουσιάζονται τα παθέματα με ορισμούς και μετά το τμήμα για την πρόθεση της συζήτησης ε, με την δυνατότητα παρουσίασης ε, της οδού που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μία δημόσια κρόση θα ήταν ιδιαίτερα θετική ιδιαίτερα όσον αφορά τα 4 και το 5 του εγγράφου που έχει παρουσιαστεί. Όσον αφορά τα πλαίσια του, της παρουσίασης του θέματος, μπορεί κανείς να τα συμμερίζεται ή όχι, αλλά είναι αξιόλογο και ακέραιο και έντιμο αυτό το οποίο εμφανίζεται σε σχέση με τα επιχειρήματα για αυτό το θέμα. Τώρα, αν τα συμμεριζόμαστε ή όχι, αυτό εξαρτάται από τις πολιτικές οικογένειες στις οποίες ανήκουμε. Και το θέμα τώρα και των κινδύνων και των ενδεχομένων μπορεί να είναι κάτι πολύ θετικό και σε σχέση με την ε, τεχνολογία και ε, τη δυνατότητα δημιουργίας ε, δυνατοτήτων ισότητας αυτό απότερα μπορεί ίσως να επιτευχθεί είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε το δίκτυο ως ένα περίπλοκο σημείο όσον αφορά την όρημη άρθρωση των επιχειρημάτων και των θεμάτων και για τις κατηγορίες που παρουσιάζονται που μπορούν να ακολουθηθούν υπάρχει μια να προσφερθούν στα πολιτικά κόμματα όλα τα μέσα ώστε υπάρχει ο κίνδυνος ε, να, και πρέπει να ληφθεί αυτός ο κίνδυνος υπόψη. Δεν είναι το ιδανικό σημείο για την ε, τοποθέτηση από αυτών των θεμάτων. Ε, Οι κίνδυνοι που ελοχεύουν πρέπει να εξεταστούν και επίσης ε, θα ήθελα να πω ότι είναι πραγματικά πολύ θελκτικό και θα έπρεπε να μπορέσουμε να διατυπώσουμε προτάσεις, διότι είναι πραγματικά έντιμος ο τρόπος αυτής της ε, παρουσίασης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Σπινέλη για την Ενωτική Αριστερά. Και, ε, Σε ευχαριστώ Ντανούτα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Χαουρέγγι για αυτό το πρώτο έγγραφο το οποίο υπέβαλε το οποίο δεν νομίζω ότι έχει ιδεολογική χρειά. Νομίζω ότι ε, φωτογραφίζει πραγματικά την υφιστάμενη κατάσταση. Η υφιστάμενη κατάσταση αντιστοιχεί σε μια κρίση της δημοκρατίας. Μολονότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμα σε πολύ αρχική φάση, συμφωνώ με τις προτάσεις που κάνει ο εισηγητής και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε μια πιο ευρεία συμμετοχή των πολιτών, ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια γενική πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, ότι θα πρέπει να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το ψηφιακό χάσμα και να προωθήσουμε τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να έχουμε όσο δυνατό μεγαλύτερη διαφάνεια. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ το ότι κάνετε μία αναφορά στο ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα. Γνωρίζουμε ότι η όλο και μεγαλύτερη χρήση των νέων αφοτεχνολογιών βάλει κατά των προσωπικών δεδομένων και τη ιδιωτική ζωή. Θα ήθελα να κάνω κάποιε πρώτε γενικέ παρατηρήσει που θα ήθελα να ενσωματωθούν στη μελλοντική εκδοχή του εγγράφου σα. Πρώτον, η ε, ανάπτυξη αυτή τη ηλεκτρονική δημοκρατία θα πρέπει να αποτελέσει μια συγκεκριμένη διαδικασία, μια προοδευτική διαδικασία προς ε, τον απότερο στόχο της ε, λήψης ε, αντιπροσωπευτικών ε, δημοκρατικών αποφάσεων, δηλαδή να μπορέσει η ηλεκτρονική αυτή δημοκρατία να λειτουργεί ακόμα και στην περίπτωση που οδηγούμεθα προς μια συγκεκριμένη λήψη αποφάσεων μέσω δημοψηφίσματος, εκλογέ, εκλογών κτλ είναι πολύ σημαντικό να μην αποτελέσει αυτό σκοπό ηλεκτρονική δημοκρατία, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση αυτή μόνο για να επικυρωθούν αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί εκ των άνω και ενδεχομένω μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επικρατήσει το status quo. Αντίθετα, θα πρέπει αυτή η ηλεκτρονική δημοκρατία να επιτρέψει να έρθουν πιο κοντά οι πολίτες με τα νέα αυτά μέσα και να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν υπέρ της δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να ευνοήσουμε κάποιες συνθήκες που να ευνοούν την ε, κοινωνική ανάπτυξη των πολιτών, οι οποίοι να μπορούν τελικά να συμμετέχουν ενεργά σε μια τέτοια δημοκρατική διαδικασία. Και ακριβώ για αυτό το λόγο νομίζω ότι στην έκθεση θα πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά και στον ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα, ο οποίος μπορεί να μας επιτρέψει να καταρρύψουμε αυτή τη στιγμή τα εμπόδια και τα φράγματα τα οποία έχουν υψωθεί στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα όσον αφορά τη ζωή των πολιτών. Δεύτερον, η ηλεκτρονική δημοκρατία νομίζω ότι αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο της ίδιας της έννοιας της δημοκρατίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο νομίζω ότι τα δικαιώματα και οι βασικές αρχές της δημοκρατίας θα πρέπει να αναγνωρίζεται και στα πλαίσια αυτής της ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Στην πράξη λοιπόν χρειαζόμαστε πάρα πολλά εχέγγυα, πάρα πολλές διασφαλίσεις οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση της πραγματικής ανάπτυξης της δημοκρατίας μέσω των νέων αυτών νέων τεχνολογικών μέσων. Θα πρέπει να Ισχύουν εδώ πέρα όλα τα εχέγγυα για την προστασία των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να σας υπενθυμίσω ότι στην Ιταλία στις 28 Ιουλίου του 2015 εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο μας μια χάρτα για τα ψηφιακά δικαιώματα, τα δικαιώματα στο διαδίκτυο. Και αναγνωρίζονται λοιπόν τέτοιες εγγύσεις στα πλαίσια της χρησιμοποίησης του διαδικτύου. Πρώτο δικαίωμα είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να εγκριθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρίτη παρατήρηση. Όπως ακριβώς λέγεται και από τον ίδιο τον εισηγητή, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε την πιο ευρεία δυνατή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όχι μόνο όσον αφορά την τεχνολογική διάχυση του νέου αυτού μέσου, αλλά όσον αφορά και κυρίως την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχει το διαδίκτυο στα πλαίσια απόλυτης διαφάνειας. Είναι σημαντικό να μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτε στι δημοκρατικέ διαδικασίε και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν έχουν τι απαραίτητε πληροφορίε και την απαραίτητη ενημέρωση. Η γνώση λοιπόν αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί κοινό καθολικό ανθρώπινο αγαθό. Και θα πρέπει να έχουμε μια καθολική πρόσβαση, ισότιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς καμία διακριτική μεταχείριση, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην κατάρριψη οποιοδήποτε εμποδίου και οποιοδήποτε περιορισμού όσον αφορά την άσκηση αυτού του δικαιώματος. Παράλληλα, αυτό θα πρέπει να δημιουργεί μια αρνητική υποχρέωση όσον αφορά τα κράτη-μέλη, δηλαδή τα κράτη-μέλη να μην θέτουν κανένα εμπόδιο όσον αφορά την πρόσβαση αυτή μέσω διαφόρων μεθόδων όπως η λογοκρισία ή άλλες μέθοδοι ε, περιορισμού στο όνομα πάντα της ασφάλειας, της εθνικής και το καθεξής. Κάποιος αναφέρθηκε σε μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε βαθιά γνώση και επιφανειακή γνώση που οδηγεί σε ένα κατακαιρματισμό όσον αφορά την γνώση στο διαδίκτυο. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την σύγκριση, με αυτή την αντιπαράθεση. Νομίζω ότι υφίσταται ακόμα και στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή μια βαθιά γνώση των πραγμάτων Απλώς δεν μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή πού ακριβώς εκφράζεται αυτή η βαθύτερη γνώση. Πολλές φορές δεν τη βλέπουμε εξαιτίας ε, των ε, κλασικών μέσων που ακόμα εξακολουθούν και χρησιμοποιούνται ή που επηρεάζονται πολύ από την οικονομική κρίση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της προώθησης προγραμμάτων e-learning, ηλεκτρονικής ε, κατάρτισης θα μπορούσε να βοηθήσει τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν περισσότερο τις νέες αυτές τεχνολογίες. Και τα προγράμματα αυτά μπορούν ήδη να αρχίσουν να εφαρμόζονται και στα σχολεία. Τέλος, προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε περισσότερο και τη συμμετοχή αλλά και τη διαφάνεια, θα πρότεινα και πρόκειται να το πράξω συγκεκριμένα και ως ασκιώδης εισηγήτρια στις επαφές που θα έχουμε στο μέλλον. Θα προτείνω λοιπόν κάποια άλλα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν σε ενωσιακό επίπεδο και θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτον, μία αναθεώρηση του κανονισμού 211 του 2011 προκειμένου να δώσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες υποχρεωτικά ένα μέσο ηλεκτρονικής συμμετοχής το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στη συνέχεια. Νομίζω ότι ε, πολλές φορές είναι εντυπωσιακή και το λέω ηρωνικά η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε φορά που ε, συγκαταβατικά απαντά σε όσους την επικρίνουν ε, για τον τρόπο που έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμή στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Αυτό το οποίο μας λέει η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να αναθεωρήσουμε το σύστημα αυτό και μου θύμισε αυτό που είχε πει ο Μάουτσετούν για τη Γαλλική Επανάσταση, ο οποίο είχε πει «It's too early to say», είναι πάρα πολύ νωρί προκειμένου να τοποθετηθώ, προκειμένου να εκφράσω μία άποψη. Σαν το Μάου Τσετούγκ μίλησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν τη γίνουν επικρίσει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Έπειτα, μία νέα πρωτοβουλία όσον αφορά του καταγγέλτε, του πληροφοριοδότε, του whistleblowers, προκειμένου να αναγνωρίζεται περισσότερο ο ρόλος τους για το δημοκρατικό έλεγχο στα πλαίσια του διαδικτύου. Τρίτη πρόταση, θα ήταν πολύ θετικό να δούμε αν μπορούμε να επεκτείνουμε περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο διάφορα, διάφορες μεθόδους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δημοψηφίσματα, περισσότερα δημοψηφίσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πασκάλ Ντιουρόν δεν είναι εδώ πέρα. Ποιος θα μιλήσει εξ ονόματος του Πασκάλ Ντιουρόν. Ναι, εσείς και μετά ο Μάξ. Σας ακούμε. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου, φίλε Χάουρικη, να ξεκινήσω με ένα θέμα. Με ενδιαφέρει το έγγραφο, με ένα γλωσσικό θέμα που θα ήθελα να σχολιάσω στα ισπανικά υποχρεωτικά επαναλάβατε δύο φορές μια φράση ότι δεν βαίνει καλώς η δημοκρατία, είπατε. Υποθέτω ότι δεν είναι πολιτικό ισχυρισμός, διότι δηλαδή να πει κανεί κάτι τέτοιο για την Ευρώπη και τη δημοκρατία, αλλά είναι κάτι θεραπευτικού χαρακτήρα, όπου δηλαδή λέμε δεν ε, βαίνει καλώς αυτή τη στιγμή, γιατί θα ήταν πραγματικά τρομερό να πει κανείς ότι η δημοκρατία χωλαίνει, ε, αναζητήσατε λοιπόν ένα μέσο που θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση της δημοκρατίας. Πολύ καλά λοιπόν και στη συνέχεια κάνατε λόγο για καθαρή πολιτική δράση, για καθαρή πολιτική δραστηριότητα αναφερόμενο σε ψηφοφορίες, διαβουλεύσεις κτλ. Και έρχομαι τώρα στο σημείο το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό εδώ για μένα και είναι το εξής. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως όταν μιλάμε για την ψηφιακή δημοκρατία. Σαν, και αυτό φαίνεται από το έγγραφο, σαν η δημοκρατία ουσιαστικά να ήταν ψηφοφορικού χαρακτήρα ή ε, για, την, για ψηφοφορίες, για διαβουλεύσεις, ε, ψηφοφορίες, ψήφιση, ενώ για τη δημοκρατία ο κύριος χαρακτήρας είναι ο κοινωνικός χαρακτήρας, κοινωνικής δημοκρατίας. Όταν ενδιαφερόμαστε για την πολιτική συμμετοχή και δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών κάνουμε κάτι θετικό, αλλά θα πρέπει προηγούμενα να ενδιαφερθούμε για κάτι άλλο. <clears throat> για την εκπαίδευση και την παιδεία την πολιτική και δημοκρατική των πολιτών. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο δεν βρίσκεται λοιπόν στο έγγραφο και απουσιάζει, ενώ θα ήθελα να βρισκόταν στο έγγραφο και να υπήρχε μία αναφορά στα μεταξύ των ε, επτά σημείων για, στο τέταρτο για παράδειγμα να γίνεται λόγος για τα κέντρα εκπαίδευσης ε, και στην ψηφιακή δημοκρατία θα έπρεπε να αναφερόμαστε στο ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει στα σχολεία, στην εκπαίδευση αυτό το στοιχείο. Και αυτό πάλι μπορεί να είναι ένα θέμα για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Αλλά μια και εξετάζουμε αυτό το θέμα σε σχέση με τα σχολεία, όταν αρχίζουν οι μαθητές να εξοικειώνονται με τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι ψηφιακού χαρακτήρα, ηλεκτρονικού χαρακτήρα και αρχίζουν να τα απορροφούν και να τα ενσωματώνουν, να τα αφομοιώνουν, και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν ακόμα κάποιες υποχρεώσεις ε, ψηφοφορικού ε, ε, πολιτικού χαρακτήρα. Πολύ θετικό αυτό λοιπόν. Θετική εκπαίδευση και εξοικείωση πριν από οποιαδήποτε ε, δράση ε, όσον αφορά τον χαρακτήρα ψηφοφοριών να εξοικειωθούν οι μαθητές ε, με αυτά τα θέματα για να υπάρχει μια ρητή αναφορά στα σχολεία και στα κέντρα ενημέρωσης των πολιτών. Έτσι λοιπόν στη συνέχεια δεν θα έρθει αυτό σαν κάτι το οποίο με κάποιο πραξικόπημα ή εξαπίνης δημιουργεί δημιουργείται και το οποίο μας ευνηδιάζει, αλλά θα έχουν προετοιμαστεί και θα έχουν εξοικειωθεί ε, διαβίου πλέον από ε, ε, μια πολύ πρώιμη φάση, νωρίς στην ηλικία τους οι πολίτες ως μαθητές. Γι' αυτό διαδραματίζει η παιδεία ένα πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να την εντάξουμε και να υπάρχει αυτή η αναφορά στην παρέμβαση. Ευχαριστώ. E Σας ευχαριστούμε κύριε Αντινόλφη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο για αυτό το έγγραφο εργασίας, το οποίο θεωρώ ότι είναι καλό. Και κυρίως σας ευχαριστώ γιατί αναφερθήκατε και στη στάση των πολιτών απέναντι στην κρίση αξιοπιστίας αυτή τη στιγμή της πολιτικής, ιδίως στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το βλέπουμε από όλα αυτά τα στατιστικά δεδομένα, από τη χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές, Ανήκω στο κόμμα Cinque Stelle, το κίνημα των πενταστέρων της Ιταλίας και όπως γνωρίζετε ορισμένοι, εμείς δημιουργηθήκαμε μέσω του διαδικτύου και χρησιμοποίησαμε πρώτα απ' όλους τις νέες αυτές τεχνολογίες. Όχι όμως για τους λόγους που ανέφερε ο κύριος Πρέντα, αλλά επειδή συνειδητοποιήσαμε ότι μέσω των νέων αυτών μέσων μπορούμε να χρησιμοποιήσουν με νέες μορφές επικοινωνίας με τον πολίτη, για να φέρουμε την πολιτική πιο κοντά στους πολίτες. Προφανώς υπάρχουν κίνδυνοι στη χρησιμοποίηση των νέων αυτών τεχνολογιών. Οι κίνδυνοι που αναφέρει και ο συνάδελφος στην έκθεσή του. Οι κίνδυνοι όμως αυτοί υφίστανται ούτως ή άλλως, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά μέσα. Για παράδειγμα, ανάμεσα στους κίνδυνους που αναφέρατε ήταν ε, και η χειραφόρων μέσων από τις συντεχνίες, από τα λόμπι. Με αυτό υφίσταται ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή. Αναφερθήκατε στην εκλογική απάτη. Με εκλογική απάτη λαμβάνει η χώρα ακόμα και αν δεν υιοθετήσουμε ηλεκτρονικά μέσα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να δούμε όλες αυτές τις αρνητικές πτυχές. Παράλληλα όμως δεν νομίζω ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ανησυχήσουμε υπερβολικά και να διστάσουμε να εγκρίνουμε νέα μέσα μόνο και μόνο επειδή ελοχεύουν κάποιοι κίνδυνοι. Όσον αφορά την εκπαιδευτική περισσότερο πτυχή, θα γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Πολιτισμού για το ζήτημα αυτό, αλλά και από προσωπική πείρα μπορώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε την πτυχή αυτή νομίζω ότι μπορεί να επιλύσει πάρα πολλά από τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε πριν από λίγο. Μάλιστα στην Επιτροπή Πολιτισμού εγκρίναμε ένα σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με τον ψηφιακό αναλφαβητισμό προκειμένου να καταφέρουμε να βοηθήσουμε όσο, όσο δυνατόν περισσότερους πολίτες να μάθουν πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τα νέα αυτά τεχνολογικά μέσα. Αν δεν υπάρξει αυτή η κατάρτιση, αν δεν υπάρξουν αυτά τα προγράμματα, προγράμματα δεν θα μπορέσει ο πολίτης να εξοικειωθεί με τα νέα αυτά μέσα. Τα προβλήματα αυτά έχουμε αρχίσει να τα βλέπουμε ήδη από τώρα. Πάρα πολλοί πολίτες που δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι εκπρόσωποι τους. Πάρα πολλοί πολίτες ε, οι οποίοι ε, μην έχοντας την απαραίτητη κατάρτιση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική, πολλές φορές λειτουργούν εντελώς παρορμητικά αν θέλουμε πραγματικά να διατηρήσουμε αυτή την καταπληκτική ευρωπαϊκή δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο διορατικοί και να καταφέρουμε με τον ένα τον άλλο τρόπο να περιορίσουμε όλες αυτές τις ακραίες πολιτικές τάσεις που βλέπουμε σε όλες τις γωνιές της Ευρώπης. Όπως σας είπα θα γνωμοδοτήσουμε στην Επιτροπή Πολιτισμού. Θα επικεντρωθούμε στις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με διάφορα προγράμματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί και θα προωθήσουμε και διάφορες δημόσιες πρωτοβουλίες ε, όπως αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας μην είναι μόνο ιδιωτικό φορέας ο πλέον αρμόδιος και για το ζήτημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε και μια πολιτική ανοιχτού ελεύθερου λογισμικού, η οποία θα προωθεί τη διεύρυνση της γνώσης και που δεν θα περιορίζεται μόνο από τις εμπορικές εφαρμογές, αν θέλετε, των νέων αυτών τεχνολογιών και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και πρέπει επίσης να πούμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε κάποια μέσα τα οποία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από διάφορες πολιτικές δυνάμεις. Κάτι ακόμα. Ένα ενδεχομένω περίεργο ή νέο μέσο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το οποίο έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται ουσιαστικά είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών που θα πρέπει νομίζω να προωθηθεί ακόμα περισσότερο. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε περισσότερο τη συμμετοχή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Μα έχουν μείνει τρει ομιλητέ, Άντερσον, Μπρέσο και Σόπλινγκ, και μετά κλείνω τον κατάλογο. Μαξ, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ. I would like to say this is very interesting. Ε, καταρχήν το έγγραφο μου φαίνεται ενδιαφέρον, κύριε Σιγητά. Έχω δύο προτάσεις και δύο σχόλια από αυτού. Πιστεύω ότι ήταν ε, εξαιρετικά χρήσιμο, αν ήταν ευκολότερο για τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών, να παρακολουθούν και να κατανοούν την νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και ε, να έχουμε έναν αντίκτυπο στη νομοθετική διαδικασία σήμερα, πρέπει να έχουμε πολύ καλές επαφές ή να πληρώσουμε ε, αποτελεσματικούς λομπίστες. Αν όμως κανείς έχει όλες τις ελευθερίες από το διαδίκτυο με εύληπτο τρόπο κατανοητό, θα ήταν πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα και θα έχει χρόνο ο κόσμος να καταλάβει και να εξοικειωθεί με την ομοθετική διαδικασία. Το δεύτερο μου σχόλιο μπορεί να είναι κάπως ε, επίμαχο, αλλά πρέπει να υποθεί. Σε ένα έγγραφο, ιδιαίτερα σε ένα έγγραφο εργασίας, για την ηλεκτρονική δημοκρατία. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουμε να πούμε κάποια λόγια για τον κίνδυνο των στρεβο... στρεβλωτικών αποτελεσμάτων που μπορεί να έχει στο κοινοβουλευτικό έργο η πληθώρα πληροφοριών στο δίκτυο. Αυτός ο πληθωρισμός πληροφοριών κάτι που κάνει τον κόσμο να προσπαθεί να ποσοτικοποιήσει κάτι που δεν επιδέχονται ποσοτικοποίηση. Αυτό ε, επηρεάζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα. Ενώ φυσικά τη βαθμολόγηση των ευρωβουλευτών, κάτι που στρεβλώνει τα μάλλον το κοινοβουλευτικό έργο. Μάλιστα σήμερα άκουσα κάποια στατιστικά στοιχεία του Ράινερ Βίλαντ που μου είπε ότι είχαμε μία αύξηση το δηλώσεων ψήφων από λιγότερο από 800 σε 60.000. Οπότε μπορεί πολλές από αυτές τις δηλώσεις ψήφου να είναι εύλογες. Οι περισσότερες όμως γίνονται μόνο και μόνο για να συγκεντρωθούν στατιστικά μόρια και να πετύχει καλύτερη κατάταξη στο σύστημα κατάταξη των βουλευτών που δημιουργεί σφαλμένες εντυπώσεις, είναι δαπανηρό και στρεβλώνει την εικόνα του Κοινοβουλίου αλλά και του κοινοβουλευτικό έργο. Αυτό το πρόβλημα δεν πρόκειται να το λύσουμε με την έκθεση Χαουρέγγια Τόντο, αλλά πιστεύω ότι χρήζει προσοχής και αυτό το πρόβλημα. Άλλο σχόλιο για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εγώ είμαι τεχνολάγνος ε, αν έχετε χρόνο αύριο το πρωί, ελάτε στο σεμινάριο για το ρομπότ, θα, τη ρομποτική που θα κάνει η Γιούρη. Αλλά το, η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι πολύ προβληματική. Γιατί έχουμε κακό σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που δεν μπορεί να εξακριβωθεί από ανεξάρτητη πηγή. Και δυστυχώς το εσθονικό σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν ε, υπόκειται σε ανεξάρτητο έλεγχο. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που διαχειρίζονται το σύστημα πρέπει να τους έχουμε εμπιστοσύνη, αλλά η ανεξάρτητη ε, δεν εξακριβώνεται ε, η κυρότητα του συστήματος από ανεξάρτητο ελεκτή. Και άρα το σύστημα είναι ευάλωτο στην εκλογική απάτη. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Και τέτοιου είδου προβλήματα θα πρέπει να αναλυθούν πιο διεξοδικά στην έκθεση, γιατί θα ήταν επικίνδυνο ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, να εκλέγεται από ένα σύστημα που είναι ευάλωτο στο, στους hacker. Στην ηλεκτρονική χειραγώγηση και άρα μπορεί να υπόκειται σε εκλογική απάτη. Τώρα, κατάχρηση πληροφοριών, χειραγώγηση από τους λομπίστες. Οι πληροφορίες που ήταν δημόσια προσιτές κυρίως χρησιμοποιούνται από επαγγελματίε λομπίστες ή ε, συντεχνιακά συμφέροντα που ε, κάτι που αντιβαίνει στο σκοπό της διαφάνειας. Είμαι Σουηδό και οφείλω να ομολογήσω την αντίθεσή μου στην προσέγγιση αυτή. Η εμπειρία που έχουμε στη Σουηδία μα έχει δείξει ότι η διαφάνεια είναι πολύ καλό πράγμα, πολύ θετικό. Και κυρίω οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί που ζητούν τι πληροφορίε και τι χρησιμοποιούν. Που σημαίνει ότι ο κόσμο έχει εμπιστοσύνη στο σύστημα. Οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι πολιτικοί κάνουν πολύ λιγότερα λάθη και πολύ λιγότερο συζητήσιμες αποφάσεις όταν γνωρίζουν ότι θα τους ελέγξουν οι δημοσιογράφοι, θα διαφερθούν οι δημοσιογράφοι και αυτό είναι θετικό γιατί δημιουργεί συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού στην πληροφόρηση. Γιατί όλοι όσοι πραγματικά θέλουν να ενημερωθούν για κάτι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τις ίδιες πληροφορίες και όχι μόνο ε, οι λομπίστες που έχουν τις καλύτερες επαφές και σχέσεις. Μπορεί να τελικά συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, αλλά σας προειδοποίησα ότι θα χρειαστεί να επανέλθουμε στο θέμα αυτό πολλές φορές. Η κυρία Μερσέντες Μπρέσο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Ραμόν για το έγγραφο αυτό εργασίας το οποίο είναι πυκνό στις προτάσεις του και πάρα πολύ σημαντική δυνατότητα να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και να σκεφτούμε λίγο περισσότερο ποια θα είναι η στάση μας για το ζήτημα αυτό. Εσύ έπειτα θα κρίνεις πώς και αν θα λάβεις υπόψη να τις παρατηρήσεις τις οποίες κάνουμε εμείς σήμερα. Το τμήμα αυτό το οποίο χαρτογραφεί την κατάσταση με βρίσκει πραγματικά σύμφωνη. Όντως έτσι έχουν τα πράγματα στη σημερινή δημοκρατία ενδεχομένως να μην ενταχθούν βέβαια όλα αυτά τα στοιχεία στην επίσημη έκθεση την οποία θα υποβάλεις, γιατί ουσιαστικά προσπαθείς αυτή τη στιγμή να μας βοηθήσεις να σκεφτούμε λίγο περισσότερο το ζήτημα για να καταλήξουμε τελικά σε ένα πιο πολιτικό κείμενο, σε ένα σύνηθες κείμενο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ θετικές οι παρατηρήσεις που γίνανε στο κείμενο αυτό και επικεντρωνόμαστε όντως περισσότερο στο ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί νομίζω ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τις νέες αυτές τεχνολογίες, τα νέα αυτά ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης. Γιατί εδώ πέρα στο ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε ακόμα πιο μακριά από τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Άρα εδώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να οργανωθούμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συνδοθούμε με όλους αυτούς τους πολίτες. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης μπορούμε να εγκρίνουμε κοινού κανόνες που θα μπορούσαν στη συνέχεια να υιοθετήσουν και τα ίδια τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανόνες βέβαια οι οποίοι δεν μπορούν σε μια πρώτη φάση να είναι δεσμευτικοί. Επομένως κάποιες κατευθύνσεις θα δώσουμε και δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε κατά τρόπο δεσμευτικό για τα κράτη-μέλη. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η διάκριση αυτή που έκανες ε, ανάμεσα στο e-governance, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση δηλαδή, το e-government, την ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση και το e-democracy, την ηλεκτρονική δημοκρατία. Όσον αφορά το e-government, την ηλεκτρονική δηλαδή δημόσια διοίκηση, συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι ε, οι νέες τεχνολογίες, τις πληροφορίες και των επικοινωνιών μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τις διοικητικές υπηρεσίες που παρέχουν τα κράτη-μέλη, από ηλική καταρχάς πλευράς, καθότι θα προβλέπεται μια ηλεκτρονική διασύνδεση, και σε προσωπικό επίπεδο, επειδή οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως τα νέα αυτά μέσα και να έχουν ένα είδος σχέσης πιο αποτελεσματική με την δημόσια διοίκηση. Θα μπορούν οι πολίτες δηλαδή να υποφελούνται των υπηρεσιών που παρέχει το δημόσιο ηλεκτρονικός. Αυτό βελτιώνει προφανώς την καθημερινή ζωή των πολιτών. Δεν νομίζω ότι κανείς αντιτίθεται στην ιδέα αυτή ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση. Το πρόβλημα έγκυται περισσότερο στη δυνατότητα πρόσβασης. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή με τις περιοχές εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ήπεθρο ή τις ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα σύνδεσης. Δεν πρέπει οι πολίτες στις περιοχές αυτές να απομονωθούν. Νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέψουμε διάφορα μέτρα υποστήριξης των πολιτών αυτών. Να υπάρχουν τουλάχιστον θα λέτε, κάποιοι φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πολίτες στις περιοχές αυτές να συνδοθούν με τη λεγόμενη ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση, χωρίς να χρειάζεται οι πολίτες αυτοί να διανύσουν ε, τεράστιες αποστάσεις προκειμένου να φτάσουν σε κάποια πόλη όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές οι υπηρεσίες. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο, χωρίς ενσύρματη σύνδεση, δηλαδή Wi-Fi, τα οποία να λειτουργούν δωρεάν. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί μόνο αν επιλύσουμε τα τεχνικά αυτά προβλήματα θα καταφέρουμε να επιλύσουμε και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία εντοπίζει η έκθεση αυτή. Αν δεν καταφέρουμε να έχουμε μια καθολική ισότιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο, τότε βαθαίνει περισσότερο το ψηφιακό χάσμα και επιδεινώνεται περισσότερο και η κατάσταση της ίδιας της δημοκρατίας. Όσον αφορά τώρα το e-governance, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα πρέπει να έχουμε ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις. Το λέτε και εσείς στην έκθεσή σας. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι αυτό είναι ουσιώδες. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες ή σε μεμονωμένα κράτη-μέλη ενδεχομένως να επηρεάζουν ένα μικρό αριθμό μόνο ενδιαφερομένων μερών και μόνο αυτοί τελικά να συμμετέχουν σε αυτές τις διαβουλεύσεις. Νομίζω ότι μέσω της ηλεκτρονικής μορφής των βρίνουμε τον αριθμό των διαφορεμένων φορέων ή ακόμα και πολιτών που συμμετέχουν στις διάφορες διαβουλεύσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο στη δικασία λήψης αποφάσεων. Μια τέτοια λοιπόν διαβούλευση, κατά την άποψή μου, η κλασική δηλαδή, είναι κάπως ψυχρή. Δηλαδή ανταποκρίνεται σε λίγους πολίτες και σε λίγους φορείς. Και ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται στο δημοκρατικό μοντέλο το οποίο θα θέλαμε. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις αλλά και για τις ηλεκτρονικές εκλογές να υπάρχει το απαραίτητο επίπεδο πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών. Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να διευθετείται μέσω αυτού που εσύ αποκαλεί στην εκθεσή σου e-governance, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στα πλαίσια λοιπόν του e-governance θα πρέπει να έχουμε πιο ευρείε διαβουλεύσει, ένα καλύτερο έλεγχο τη ποιότητα, αν πραγματικά ενημερώνονται ισότιμα όλοι οι πολίτε, αν όντω έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί πολίτε δεν είναι παρκώ ενημερωμένοι και χάνουν πάρα πολλέ ευκαιρίε που του δίνουν αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήγουν να λένε μετά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί με διαφάνεια. Και το πιο πολύπλοκο για μένα κεφάλαιο είναι περισσότερο αυτό της e-democracy, της ηλεκτρονικής δημοκρατίας. Εδώ πέρα έχουμε τις κλασικές μεθόδους, αν θέλετε, των εκλογών, του δημοψηφίσματος και το καθεξής για κάποια όμως ζητήματα τα οποία είναι τους άλλους δεδομένα, για τις πιο κλασικές μορφές εκλογών αν θέλετε. Νομίζω ότι με τα νέα αυτά μέσα μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο την ιδέα της ανοιχτής συμμετοχικής δημοκρατίας, όπως στην περίπτωση του Πόρτο Αλέγκρε, όπου ξέρετε ότι πάρα πάρα πολλοί πολίτες είχαν ε, συμμετάσχει. Προφανώς δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αλλά θέλουμε να έχουμε επιπλέον μέσα τα οποία να πλαισιώνουν, να συνοδεύουν την πιο κλασική μορφή της δημοκρατίας. Θέλουμε και τα νέα αυτά μέσα όμως να είναι σωστά οργανωμένα και διαρθρωμένα. Και ακριβώς αυτό το ζήτημα της διάρθρωσης των νέων δημοκρατικών ηλεκτρονικών διαδικασιών όπως ε, ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα κτλ. πρέπει να μας απασχολήσει. Πρέπει και εκεί να έχουμε τα απαραίτητα χέγγια, τι απαραίτητε εγγυήσεις ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη ενημέρωση και το καθεξής. Πρέπει λοιπόν επ' αυτό να εργαστούμε ακόμα πολύ. Συμφωνώ πάντως ε, με τη συνάδελφο που είπε πριν από λίγο ότι δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τα σφάλματα που ενδεχομένω να έχουμε κάνει ή να προκύψουν. Ανταυτού νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε τα απαραίτητα μέσα δημοκρατικής συμμετοχής, τα οποία θα εγγυώνται την ποιότητα, αν θέλετε, της δημοκρατικής αυτής συμμετοχής. Χαρακτηριστικό της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, υπάρχει ένα συγκεκριμένο εκλογικό σώμα, εκλέγουν οι πολίτες αυτόν που θα τους εκπροσωπήσει, ο οποίος τη συνέρχεται σε επαφή ή ελέγχει την εκτελεστική εξουσία, αλλά υπάρχουν παράλληλα για το σύστημα αυτό συντάγματα τα οποία πραγματικά διαρθρώνουν αυτή τη μορφή δημοκρατίας. Η ιδέα η παράλληλη της δημοκρατικής ηλεκτρονικής συμμετοχής παραμένει πιο ασαφής αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν αυτή να καταφέρουμε να τη διαρθρώσουμε με ένα πιο συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν θεσπίσουμε κανόνες. Κανόνες όσον αφορά την καθολική πρόσβαση. Κανόνες όσον αφορά τη γνήσια συμμετοχή των πολιτών και όχι τη χειραγώγηση των νέων αυτών μορφών δημοκρατίας. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια συμμετοχική δημοκρατία η οποία θα είναι γνήσια και η οποία τελικά δεν θα αποτελεί αντικείμενο χειραγώγησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο τελικά στην όλη αυτή η ιστορία. Αυτή τη στιγμή θα υπάρχουν αυτά τα νέα μέσα δημοκρατικής ηλεκτρονικής συμμετοχής, θα θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν και οι ίδιοι οι πολίτες. Θα καταφέρουμε να αυξήσουμε την συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και θα υπάρχουν περισσότερες διευκολύνσεις προκειμένου να συμμετέχουν οι πολίτες ενεργά στην πολιτική, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν σε κάποια άλλη πόλη, χωρίς να πρέπει να καταβάλουν άλλες προσπάθειες να ξεπεράσουν κάποια εφιστάμενα εμπόδια. Όλα αυτά επιλύονται με μια σωστή χρήση των νέων αυτών ηλεκτρονικών μέσων συμμετοχικής δημοκρατίας. Βλέπω όμω του μορφασμού που κάνει αυτή τη στιγμή η πρόεδρο, η οποία προφανώ θέλει να ολοκληρώσει την παρέμβασή μου. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστούμε πολύ και για την παρέμβαση που ε, ίσως θα μπορούσε να είναι πιο σύντομη. Θα είμαι πολύ σύντομος, πραγματικά πολύ σύντομος. Να επανέλθω στην προηγούμενη παρέμβαση που θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και έχετε δίκιο για την ποσοστοποίηση του μη μετρήσιμο, του μη καθορίσιμου και ε, σε σχέση με έναν αλγόριθμο που θα μπορούσαν διαφορετικά στοιχεία να εισαχθούν ώστε να αντανακλάται η πραγματικότητα στα όσα κάνουμε με πιο επιτυχή τρόπο. Και σε σχέση με το επίπεδο, υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης για την Εσθονία δεν ε, είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι μια αναγκαία προϋπόθεση εκ προημίου ώστε να μπορεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία να λειτουργεί. Και αν μπορώ να πω κάτι στην Μπάρμπαρα ε, Σπινέλη, δεν είναι ε, αυτό που είπατε ότι είναι υπερβολικά πρόημο να κρίνει κανείς. Θα θυμόσαστε, ο Κίσιντζερ είπε ότι ήταν ο Μάρξ Ας το αφήσουμε ίσως αυτό με, εσείς ε, είχατε την ευκαιρία να το ε, γνωρίζετε αυτό. Απλά και μόνο αυτό που θέλω να πω είναι ότι ε, αν διαβάσετε είναι πολύ πιο περίπλοκη, πολύ πιο σύνθετη προσωπικότητα από τον ΜΑΟ. Σε πολλά σημεία Μπορεί κανείς να ε, γνωρίζει ότι η σημερινή ε, επικαιρότητα είναι η σημερινή ημέρα, είναι η μέρα των ευρωπαϊκών ε, δημοψηφισμάτων, η πρωτοβουλίων των πολιτών. Και είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο αναφέρθηκε. Πρόκειται για το αδικαιώμα των ίδιων των πολιτών εδώ. Η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε με αυτό είναι ένα πραγματικά λένε πολύ νεόδμητο ε, καινοφανές στοιχείο. Ε, ωστόσο αυτό σε σχέση με το έγγραφο εργασίας ε, παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να προβληματιστούμε από αυτόν. Αυτά τα οποία θα να, μπορείτε να ενθυμηθείτε για τη δική μου έκθεση για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών στο ψηφιακό επίπεδο, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Περί αυτού επρόκειτο. Ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο αυτό για το οποίο κάνουμε λόγο είναι ο συσχετισμός των πολιτών με την εξουσία. Πώς μπορεί να διαρθωθεί, να δομηθεί αυτή η σχέση και εδώ μια πρόσθετη σκέψη, το ψηφιακό θεματολόγιο, το ψηφιακό μέλλον. Τα πράγματα έχουν ήδη αλλάξει και έχουν τροποποιηθεί όλες ε, οι ε, ε, επαναληπτικές αυτές διαδικασίες γίνονται από ρομπότ και από, με μηχανικό τρόπο. Και πολύ, πολύ σύντομα ένας μεγάλος αριθμός δικηγόρων δεν θα έχουν πλέον απασχόληση ε, και μπορούμε να δούμε και σε σχέση και με τα επαγγέλματα περίθαλψης, ε, ε, ιατρικής περίθαλψης, το μέλλον και οι προοπτικές ε, πραγματικά το πώς διαγράφονται μπορεί να μας ανησυχήσουν ίσως ο τρόπος ε, με τον οποίο πρέπει να ε, δούμε αυτές τις εξελίξεις ε, εκεί όπου η ψηφιοποίηση είχε σημαντικότατες επιπτώσεις αυτά που απορρέουν από αυτή την κατάσταση εγώ δεν πιστεύω στην ιστορική αναγκαιότητα και στην ιστορική νομοτέλεια και σε σχέση με την ε, ψηφιακή εξέλιξη των πραγμάτων δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ε, αυτοεξαίρεση και θα προσέθετα δύο ή δυόμιση ακόμα επιχειρήματα θα χρειαστούμε πάρα πολλούς ειδικού, πολύ περισσότερους ειδικού για τις τεχνολογίες ε, της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας και δεν είναι όλοι πρικισμένοι και ικανοί γι' αυτό. Και δεύτερον, με θέλει ιδιαίτερα ότι η νεότερη γενεά που αυτή τη στιγμή ε, δρά προς αυτή την, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, έχει ως δεύτερη φύση το ψηφιακό ε, στοιχείο. Και ενώ έχουν ε, αυτό το, αυτά τα χαρακτηριστικά, βλέπουμε ποια είναι η δημογραφική εξέλιξη της κοινωνίας μας. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ε, ε, μια βοήθεια, μια υποστήριξη για την ε, διαβίβαση αυτών των στοιχείων για να μπορέσουν ε, να διατηρήσουν αυτή την αυτονομία στη δράση τους οι πολίτες ε, πρέπει να γίνουν πολλές προσπάθειες και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η τεχνογνωσία και η μεταφορά της είναι δαπανηρή διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Το ελέγξα και ήταν ο που το είπε αυτό. Ναι. to hear Χαίρομαι ιδιαίτερως, επιτέλους έλαμψε η αλήθεια. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι επειδή είναι ΕΛΚ. Όλοι γίναμε κομμουνιστές εδώ πέρα. Ολοκληρώσαμε με τους ομιλητές. Ίσως να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μας τον Ραμόν. Πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι παρεμβάσει που ακούστηκαν και θα εμπλουτίσουν σίγουρα το έγγραφό μου. Και δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες τώρα, διότι θα ανάλωνε πολύ χρόνο και δεν έχουμε αυτό το χρόνο στη διάθεσή μας. Ήταν ε, σε υψηλό επίπεδο η συζήτηση που διεξήχθη και πραγματικά υψηλή ποιότητας ε, και θα προσπαθήσω με αναδιατύπωση του εγγράφου δεύτερη αναδιατύπωση να προχωρήσω. Θα μπορούσαμε να είχαμε και μια ακρόαση. Έχουμε ήδη μια ακρόαση που κάναμε στο παρελθόν με κάποιους επαΐοντες για αυτό το θέμα. Μπορούμε να φέρουμε κι άλλους ακόμα επαΐοντες και να γίνει κάτι τέτοιο ως ακρόαση από πλευράς μου είμαι ανοιχτό σε κάποια τέτοια πρόταση της Προεδρίας αλλά πρέπει να εξειδικεύσουμε κάπως περισσότερο διότι αυτός είναι ο ορισμός τον οποίο ζήτησαν οι συνάδελφοι, να εξειδικεύσουμε περισσότερο και σε σχέση με κάποιες επεξηγήσεις να έχουμε τις αιτιολογικές σκέψεις και αιτιολογικές αναφορές σε σχέση με τις ιδέες που προσπάθησα να σας παρουσιάσω. Θα προσπαθήσω να το κάνω και ίσως μπορούμε να το κάνουμε αυτό και σε σχέση με μια συνάντηση με αυτό το έγγραφο. Σας ευχαριστούμε Ραμόν. Η πρόταση λοιπόν είναι ότι κατά τα τέλη του Μαΐου θα μπορούσαμε να είχαμε την επόμενη συνάντηση της Επιτροπής μας και να έχουμε μια ακόλουθη, μια επακόλουθη ανταλλαγή απόψεων και στο μεσοδιάστημα θα μπορούσατε να προετοιμάσετε, να ετοιμάσετε κάτι που θα συμπεριλάμβανε και κάποια σχόλια από τη σημερινή συζήτηση και στις 15 Ιουνίου θα έχουμε την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης 1η Ιουλίου η ιουλιου η εκνοη της προθεσμίας για κατάθεση τροπολογιών και θα τις εξετάσουμε στη συνέχεια και θα ψηφίσουμε τον όχι το Φεβρουάριο, το Σεπτέμβριο και μετά θα, θα εξεταστούν στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Εντάξει, λοιπόν, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που προτείνουμε. Κατανοώ ότι είναι πρόθυμος και ανοιχτός στα σχόλια και παρατηρήσεις που θα ήθελαν να κάνουν οι συνάδελφοι προς το Ραμόν. Τώρα, για τρία λεπτά να σας ενημερώσω για τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τους συντονιστές σήμερα. Οι συντονιστές λοιπόν αποφάσισαν να αναθέσουν τη γνωμοδότηση προς την Τζούρι για την εφαρμογή του, την για την εφαρμογή του δικαίου για το 2014, άνεμα, CNF, τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και την έκθεσή της για το ρόλο των πληροφοριοδοτών στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων, ο κύριος Μέσεριτς από το ECR. Ε, εξετάσαμε και το θέμα της ομάδας εργασίας ε, για την ερμηνεία και εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία. Ε, θα συμπροεδρεύσουν η ΑΦΚΟ και η Ε, θα συνεδριάζει απαξ το μήνα και αποφασίσαμε να συμμετέχουν εκεί και ηγητές και των δύο επιτροπών άρθρο 55 συνεργασία των δύο επιτροπών νομικών υποθέσεων και σταγματικών υποθέσεων. Μάλιστα, έχουμε και ένα πολύ ισχυρό διοικητικό επιτελείο που συνεπικουρεί ε, τα μέλη της ομάδας εργασίας. Εξετάσαμε την ανάγκη αναβολής ε, της προβλεπόμενης ε, ακρόασης 11 και 12 Ιουλίου για τις πιθανές συνέπειες των ποινικά ζητήματα. Προτιμήσαμε τον Ιούλιο να εξετάσουμε τα αποτελέσματα του Βρετανικού δημοψηφίσματος και να επανέλθουμε μετά τις χθερινές διακοπές ε, στην ακρόαση και να τη διοργανώσουμε. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι στα πλαίσια της απόφασης για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ε, των εκθέσεων ε, εφαρμογής που αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων, αποφασίσαμε ότι θα ζητήσουμε επίσημα την άδεια για να εκπονήσουμε δύο εκθέσει εφαρμογή που ήδη είχαμε αποφασίσει τον Οκτώβριο στην Επιτροπή μα και μπορούμε επιτέλου να ξεκινήσουμε τι σχετικέ εργασίε. Έκθεση εφαρμογή ε, με θέμα την εφαρμογή των διατάξεων των συνθηκών για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ο Πάολο Ρανζέλ ανέλαβε την έκθεση από το ΕΛΚ και η δεύτερη έκθεση είναι τη Μπάρμπαρα Σπινέλη με θέμα την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο. Συμφωνήσαμε για τις αυτές εκθέσεις. Ε, για τις εκθέσεις εφαρμογής ε, θα έχουμε παραλίλει το πολύ τρεις εκθέσεις και συμφωνήσαμε να τηρήσουμε τον κανόνα, δηλαδή ε, το 12 να είναι η περίοδος όπως προβλέπει ο κανονισμός για τη διεκπαιρέωση της έκθεσης, της κάθε έκθεσης εφαρμογής μέσα σε ένα χρόνο πρέπει να ολοκληρώνεται το θέμα. Σε ό,τι αφορά το, την γνωμοδότηση ε, και τον προϋπολογισμό του 2017, πρόκειται για μια ειδική διαδικασία. Συμφωνήσαμε να καταθέσουμε τις τροπολογίες για τον προϋπολογισμό μόνο στα αγγλικά, με προθεσμία την 6η Ιουνίου, γιατί την τελευταία διετία η διαδικασία δεν μας επιτρέπει να ακολουθήσουμε τις συνηθισμένες πρακτικές και πρέπει τη γνωμοδότησή μας να την υιοθετήσουμε στη συνεδρίαση του Ιουλίου. Οι τροπολογίες για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να κατατεθούν στην Ολομέλεια μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Και ήδη έχουμε αναθέσει τον Γιώργη Τσέπλιν, τον εισηγητή, να προσαρμόσει τις ε, τροπολογίες μας για τον προϋπολογισμό στη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού αν είναι θέμα χρονοδιαγράμματος, γιατί η θέση του Συμβουλίου θα υποβληθεί ε, αρκετά αργά, οπότε θα προλάβουμε να έχουμε ε, κανονική συνεδρία της Επιτροπή, οπότε θα τον αναλάβει ο συγγητής. Αυτά ως προς αποφάσει των συντονιστών. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι γίνονται δεκτές. Και περάμε στο τελευταίο σημείο τη της διάταξη. Μια στιγμή να το βρω. Είναι η γνωμοδότηση του κυρίου Γεώργη Σέπφλιν με θέμα τη δημιουργία ενός ενωσιακού μηχανισμού για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο Γιώργης είναι σε μια εκτενή γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών που είναι αρμόδια κατ' ουσία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήταν ε, ε, πολύ αγαστή και εκτενή συνεργασία που είχαμε με τη Σοφή Ίντφελτ, την εισηγήτρια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ήταν αναρρύθμιτες συναντήσεις που είχαμε, 6-7, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οι περισσότερο στο Στρασβούργο και κανένα δυο έγιναν και στις Βρυξέλλες. Η έκθεση Ίντβελτ ε, είναι έτοιμη. Και αυτό που κάνει η συγγήτρια, και εκεί θα ενταχθεί και η δική μου γνωμοδότηση, είναι να προτείνει μια διοργανική συμφωνία για να διασφαλιστεί συγχρονισμός των τριών μηχανισμών. Οι τρεις μηχανισμοί είναι της διακυβέρνησης, ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε τις 11 Μαρτίου του 2015 από, τον από την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ και που ισχύει στην περίοδο ε, για την Πολωνία, για το κράτος δικαίου. Και το Συμβούλιο, χάρη στην Ιταλική Προεδρία, έχει ένα σύστημα ε, ελέγχου μοτίμων, εξολόγηση μοτίμων, κάποιες συζητήσεις ε, διάφορες για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και η Ολλανδική Προεδρία είναι αρκετά δραστήρια ως προς το θέμα αυτό. Ένα από τα σχόλια που υπέβαλα στη Σοφία Ιντβελτ ήταν ότι καλό θα ήταν και οι τρεις μηχανισμοί να συμβαδίζουν. Εξού και η πρόταση για διοργανική συμφωνία. Γιατί όντως αυτοί οι τρεις μηχανισμοί, δημοκρατίας, κράτους δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων, μοιάζουν. Επίση προτείνει η κυρία Ιντβέλτ ένα συμβούλιο αξιολογητών για την παρακολούθηση της διαδικασίας και ένα πίνακα βαθμολόγησης επιδόσεων. Διαβάστε την έκθεση Intveld, θα δείτε πολλές φορές τα αρχικά DRF, Δημοκρατία, Κράτος Δικαίου και Θεμελιώδη Δικαιώματα. Τώρα, η δική μου γνωμοδότηση απαρτίζεται από διάφορα σημεία. Όποιο μηχανισμό και διαλέξουμε θα πρέπει να είναι δίκαιος και να εφαρμόζεται εξίσου σε όλα τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει να έχουμε διπλά μέτρα και σταθμά, ούτε να χρησιμοποιείται ο μηχανισμό ω εργαλείο μόνο ει βάρο ενό κράτου μέρου. Επίση, χρειάζεται νομική βάση. Δεν έχει νομική βάση ο μηχανισμό και το πλαίσιο τη Επιτροπή ε, δεν έχει νομική βάση. Η μόνη νομική βάση που έχουμε είναι για τις διαδικασίες επί παραβάση και το άρθρο 7. Και γι' αυτό έγινε και όλη η φασαρία. Θα θυμάστε την έκκληση των τεσσάρων υπουργών εξωτερικών πριν από λίγα χρόνια, που είπε ότι θα είναι μεταβατικός μηχανισμός, ενδιάμεσος, αλλά στερείται νομικής βάσης και το Συμβούλιο το αποσαφήνισε. Κάτι που σημαίνει όχι σήμερα, όχι αύριο, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση των συνθηκών για να δημιουργηθεί νομική βάση. Κάτι που δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο να συγχρονίσουμε τους τρεις μηχανισμούς. Η αναθεώρηση των συνθηκών για να δημιουργηθεί νομική βάση, ούτε και αυτό θα είναι εύκολο. Δεν χρειάζεται να σας κουράσω με λεπτομέρειες. Και το πρώτο τελευταίο μου σχόλιο, είναι σημαντικό να μην γίνει πολιτικοποίηση των μηχανισμών. Είναι πολύ λεπτό το θέμα και πολύ ευαίσθητο. Θα πρέπει να μείνει μακριά από πολιτικοποίηση, γιατί αν θεωρηθεί πολιτικοποιημένος ο μηχανισμός, θα θυγεί η αξιοπιστία του. Θα απαξιωθεί. Οπότε σωστό είναι να κρατήσουμε αυτή τη διάκριση. 81 τροπολογίες υπευλήθησαν, πολύ ε, χρήσιμες μερικές. Σας ευχαριστώ πάντως Βέβαια, μερικές είναι εκτός θέματος. Ε, περισσότερο αφορούν την έκθεση της κυρίας Σίντβελτ παρά τη δική μου γνωμοδότηση. Και όσοι παρακολουθούν το θέμα, παρακαλώ να υποβάλουν τροπολογίες και στην έκθεση της Σοφή Ίντβελτ. Πολύ σύντομα θα οργανώσω και συνάντηση των σχεδόν εισηγητών για να συζητήσουμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και σας ευχαριστώ θερμά γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον το εγχείρημα. Για μένα σίγουρα πάντως γιατί έμαθα πολλά αυτό. Ευχαριστώ. Ο Πέτρο Σίλβα Περέρα από τους Σοσιαλιστές τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Σεφλίν για το έργο που επετέλεσε και επίσης για την προθυμία του που δείχνει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να βρούμε λύσεις με συμβιβασμούς, διευρυμένους συμβιβασμούς. Νομίζω ότι η πρώτη αναφορά που έγινε σε σχέση με μία άρθρωση, συνεργασία με την ΛΥΜΠΕ είναι μεγάλη μεγάλης και αυτή η ιδέα για μια διαθεσμική συμφωνία για να συντονιστούν τα διαθέσιμα όργανα σε σχέση με αυτό το θέμα για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα θεωρώ ότι είναι μια καλή λύση και βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι μια λύση που έχει πολύ μεγάλο δυναμικό. Κατατέθηκαν πολλές τροπολογίες είναι η αλήθεια και καταγράφουμε αυτό σε σχέση με την διαθεσιμότητα επικοδομητικού πνεύματος συνεργασία, προθυμία συνεργασίας με επικοδομητικό πνεύμα. Επίσης ε, για τις προτάσεις που κατατέθηκαν από την ομάδα μας ε, το ίδιο ισχύει. Θα ήθελα να τονίσω δύο ή τρεις πτυχές εδώ. Πρώτα, το γεγονός ότι παρόλα τα αυτά ο μηχανισμός που έθεσε σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάπως προληπτικά ή ως πρόνοια για την ε, λειτουργικότητα επίπεδο είναι ένα σημαντικό μέσο και στο τέλος τέλος ε, αυτό εφαρμόζεται στις πιο επίμαχες περιπτώσεις ε, σε σχέση με τα θέματα που βρίσκονται υποσυζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και Έχουμε προτάσεις που έχουν κατατεθεί με αναφορές σε αυτό το μέσο που πρέπει να αξιοποιηθούν, να αναβαθμιστούν έτσι. Από την άλλη πλευρά έχουμε μία αναφορά σε τροποποίηση συνθήκων που θεωρούμε ότι μπορεί να έχει κάποιο νόημα σε σχέση με το πνεύμα το οποίο εμπνέει τον ε, εισηγητή. Δεν είναι όμως τόσο επιτακτική ανάγκη αυτή η τροποποίηση των συνθήκων, θεωρούμε εμείς. Είναι χωρίς αμφιβολία ένα νέο μέσο το οποίο εδώ ε, συνεπάγεται ένα νέο πλαίσιο σε σχέση με το να επικαλεστούμε μια τροποποίηση των συνθήκων. Γίνεται λόγος εδώ λοιπόν για ένα συμπληρωματικό στοιχείο, ένα συμπληρωματικό μέσο πρόληψης ή πρόνοιας σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 και ίσως αυτό θα μπορούσε να αποφευθεί. Δεν θα πρέπει να συρρυκνωθεί η συζήτησή μας απλά και μόνο στην τροποποίηση, μελλοντική τροποποίηση των συνθήκων, διότι θα πρέπει να δούμε ότι αυτό σε σχέση με τον χρονορίζοντα τον άμεσο δεν θα έχει κάποιες επιπτώσεις, μια και είναι πολύ πιο μακροπρόθεσμο εγχείρημα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τη σημαντική αναφορά σε σχέση με το έργο που μπορεί να αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον με μια ετήσια συζήτηση που θα διεξάγεται για αυτά τα θέματα με τη θέσπιση benchmarks βέλτιστων προδιαγραφών στοιχείων πλαισίου δηλαδή αναφοράς και αυτό θα έδινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ικανότητα, ένα μέσο επιπρόσθετο με μια πρόσθετη αξία που θα δημιουργούσαμε σε σχέση με το σημερινό πλαίσιο που ισχύει σήμερα. Αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία απορρέουν από τις προτάσεις μας και θα έλεγα ότι είναι οι πιο ουσιώδεις πτυχές αυτές και <clears throat> δεχόμεθα τις προτάσεις του εισηγητή να επικεντρώσουμε τις δράσεις μας στην πρωτοβουλία της ΛΥΜΕ, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, διότι πολλά από αυτά τα θέματα αυτά εκεί θα αναπτυχθούν και θα αναλυθούν και έτσι λοιπόν προσβλέπω στην επόμενη συνάντηση σχεδόν εισηγητών για να υπάρξει η συνέχεια αυτής της εργασίας να καταλήξουμε σε αίσιο πέρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καζίμιες Ουγιασδόφσκι. Ευχαριστώ θερμότατα τον κύριο Σέπλιν για την εκπόνηση της γνωμοδότησής του. Έχουμε εδώ διαφορετικά θέματα που είναι ελεύθερα αλλά ξεχωριστά παρόλα αυτά. Έχουμε την έκθεση της κυρίας Σόφη Ιντβελτ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Μάλιστα τον τελευταίο καιρό έχει κάνει μεγάλη στροφή η κυρία Ιντβελτ γιατί αρχικά είχε προτείνει την υιοθέτηση ενός νέου συμφώνου που θα αποτελέσει τη βάση του μηχανισμού του ελέγχου του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και μάλιστα κάποιες τροπολογίες από ευρωβουλευτές αναφέρονται σε αυτό το θέμα της ε, ε, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών ενό νέου συμφώνου για, τη για τον έλεγχο τη Δημοκρατία και του Κράτου δικαίου. Τη σύναψη τέτοιου συμφώνου από τα κράτη-μέλη. Και μετά άλλαξε αυτή την πρόταση με την πρόταση για τη διοργανική συμφωνία, που είναι μια διαφορετική μορφή ελέγχου. Εγώ πιστεύω πάντως ότι δεν στηρίζεται στις συνθήκες η πρόταση κυρία Σίντελτ. Δεν έχει βάση συνταγματική, δεν έχει βάση τις συνθήκε Γιατί μπορούμε για το εφνομοθετή να, να προβλέπουμε οργανική συμφωνία, γιατί μιλούμε για τη σχέση των θεσμικών οργάνων, αλλά δύσκολο να δεχτούμε τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας που θα έχει συνέπειες στον έξω κόσμο. Δηλαδή στα κράτη-μέλη και όχι στη σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Εγώ βέβαια δεν θέλω να αμελήσουμε το θέμα του κράτους δικαίου και είμαι υπέρ του σεβασμού του κράτους δικαίου. Γιατί νομίζω ότι θα, όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα θα ξέρουν ότι εγώ πρότεινα συμβαστική λύση για να επιληθεί το ζήτημα με το συνταγματικό δικαστήριο στην Πολωνία. Είμαι λοιπόν υπέρ της μέρημνας του, του σεβασμού του κράτους δικαίου, αλλά προσοχή. Δεν θα πρέπει ε, να προβλέψουμε νέους μηχανισμούς ελέγχου του κράτους δικαίου που δεν θα έχουν θεμέλιο τη συνθήκη. Πάντως είναι θετική γνωμοδότηση του κυρίου Σέπλινγκ. Περιέχει κάποιες προτάσεις που μας επαναφέρουν στον δρόμο της νομιμότητας. Κάτι που στερούνταν η έκθεση Υποβάλλει διαφορετική θεσμική πρόταση για τον έλεγχο. Ο κύριος Σέμπλινγκ μιλάει για συμφωνία μεταξύ των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των εθνικών κοινοβουλίων. Αυτή είναι η ιδέα που ανέπτυξε και στο έγγραφο εργασίας ο κ. Σόπλινγκ και μίλησε για προαιρετικές ετήσιες διασκέψεις με θέματα τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αυτό είναι δυνατό, γιατί προϋποθέτει συμφωνία των κοινοτικών θεσμικών οργάνων με τα εθνικά κοινοβούλια. Πάντως, επαναλαμβάνω, η, έκθεση της, η πρόταση κυρία Σίντβελτ στερείται ε, νομικής βάσης της συνθήκες. Γιατί είναι αδύνατο μια απλή διοργανική συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να έχει αποτελέσματα στις χώρες μέλη. Πάντω η γνωμοδότηση του κ. Σέπλινγκ είναι πολύ θετική και την εκτιμώ ιδιαίτερω γιατί μα επαναφέρει στο δρόμο του σεβασμού τη νομιμότητα και του σεβασμού των συνθηκών. Και στο δρόμο τη αμεροληψία και τη μη πολιτικοποίηση ε, και τη πολιτική αντικειμενικότητα και όχι τη πολιτική μεροληψία που χαρακτηρίζει την έκθεση Ιντφελτ. Επαναλαμβάνω λοιπόν εκτιμώ ιδιαίτερα στη γνωμοδότηση Σέπλινγκ, ακριβώς επειδή εκφράζει το σεβασμό στην ε, ένομη τάξη που δημιουργούν οι συνθήκες. Και προτείνει δυνατούς με βάση τη συνθήκη ε, τρόπους ελέγχου και μηχανισμούς. Σε αντίθεση με την κυρία Ιντβελτ. Η κυρία Πορτοντούα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, και εμείς επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για το έργο που επετέλεσε, διότι καταβάλει μέγιστη προσπάθεια και για τα θέματα αυτά μπορούμε πολλά να μάθουμε νομίζω σε σχέση με τη διαδικασία της ε, ε, διαβούλευσης και της ε, έκφρασης της νομοδότησης από πλευράς μας. Έχουμε το θέμα των τροπολογιών και σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο προλαλής σας. Ωστόσο, συμμεριζόμαστε ένα κοινό μέλημα, την μη πολιτικοποίηση και την αντικειμενική εξέταση αυτών που πρέπει να είναι θέματα ελέγχου, που είναι τόσο μεγάλη εμβέλειά τους για να διασφαλίσουμε ότι οι δημοκρατίες μας, τα δημοκρατικά καθεστώτα μας θα αξίζουν το όνομα δημοκρατικών καθεστώτων σύμφωνα και με το δεύτερο άρθρο της Συνθήκης Ένωσης και να εξετάσουμε τους σκόπιμους μηχανισμούς, θεσμικούς μηχανισμούς με τους οποίους μπορούμε να εργαστούμε και όσα ανέφερε ο κύριος Σέφλιν ε, όχι αποκλειστικά με την τροποποίηση των συνθήκων που είναι άλλο μέσο, να έχουμε λοιπόν μέσα δεσμευτικά μέσα υποχρεωτικής εφαρμογής να έχουμε αντικειμενικά στοιχεία ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα των δημοκρατικών καθεστώτων μας και των ελέγχων που θα διασφαλίζονται από αυτά τα καθεστώτα και που δεν έχουν προχωρήσει ίσως επαρκώς. Θα έχουμε και ευκαιρία να συνεργαστούμε με τον, με εισηγητή και ε, βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν και τροποποιήσεις, τροπολογίες σε σχέση με τη γνωμοδότηση. Είναι ένα θέμα που μας παθιάζει αυτό. Είμαι νέα ευρωβουλευτής, αλλά πολλά έχω να μάθω και να εξοικειωθώ με αυτά. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στα οποία μπορούμε να αποδηθούμε και να εργαστούμε επ' αυτών και οι αξίες αυτές και όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να μας κάνουν να ενδιαφερθούμε και να καταθέσουμε προτάσεις. Ευχαριστώ. Ο Κώστας δεν παρίσταται. Ο Greens, Από τους πρασίνους. Καμπράς παρακαλώ. Κύριε Μετσία. Uh, just to... Θα είμαι πολύ σύντομος να κάνω δύο-τρία σχόλια. Δύο-τρία σχόλια θα κάνω μόνο. Νομίζω ότι υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία και συνένεση ως προς το ότι αν δούμε τα κριτήρια της Κοπεχάγης πρέπει αυτά να τηρούνται από όλα τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές αυτές είναι ξεκάθαρες. Δεν έχουμε όμως μηχανισμούς συμμόρφωσης. Αυτό λείπει. Εκεί έγκυται το ζήτημα. Δεύτερον, όσον αφορά την νομική βάση. Ως προς αυτό δεν προβλέπεται γενική αρμοδιότητα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ωστόσο, νομίζω ότι απαιτείται απλώς πολιτική βούληση. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που δημιουργήθηκε απουσία συγκεκριμένης αρμοδιότητας και νομική του βάση είναι το άρθρο 3, 4, 5, 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να βασιστούμε στην υφιστάμενη συνένεση και πρέπει να επιδείξουμε και την απαραίτητη πολιτική βούληση που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε κάτι πολύ σημαντικό όπως πετύχαμε και με τη θέσπιση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Μάσιμο Καστάλντο δεν είναι στην αίθουσα, ούτε ο Γκέρολφ Ανενμάνσα δεν είναι εδώ, δεν νομίζω ότι θα τους αντικαταστήσει κάποιος. Υπάρχει κάποιος που θα θέλει τώρα να πάρει το λόγο. Γιώργη, ενδεχομένω εσύ να θες να ξαναπάρεις το λόγο, παρακαλώ. Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες στη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ αν δεν συμβεί τίποτα άλλο θα ψηφίσουμε στις 30 Μαΐου. Θα δώσουμε επίτα τη γνωμοδότησή μας στη ΛΥΜΠΕ και η ΛΥΜΠΕ αν δεν κάνω λάθος θα ψηφίσει στη συνέχεια στις 30 Ιουνίου. Έχουμε λοιπόν ακόμα χρόνο μπροστά μας. Αυτό ήταν ε, το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Στα διάφορα, στο σημείο 12, να σας πω απλώς ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 30 Μαΐου για μισή μέρα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγη τη συνεδρίαση. Η πρόεδρο ευχαριστεί τους δερμηνεί.